Okay, colleagues, I think we can make a start. We have an, an empty room this afternoon, but I think you will agree that... Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω η πρωινή μας ε, συνάντηση με τους προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν ε, πολύ επιτυχημένη. Είχαμε εκπροσώπους από 24 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από διάφορες χώρες της Αφρικής Νομίζω ήταν χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Αλλά ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας και να συζητήσουμε την ημερησία μα διάταξη, σημείο 12, ενίσχυση τη βιωσιμότητα του χρέου των αναπτυσσόμενων χωρών. Εγώ θυμάμαι ε, το 2000 την εκστρατεία του επιλή με την οποία είχαμε προσπαθήσει να πιέσουμε για τη διαγραφή του χρέους διαφορών αναπτυσσόμενων κρατών όμως, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και με τις πολιτικές που ακολουθούσαν τότε ε, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα διάφορα κράτη είχαν πρόσβαση σε φτηνά δάνεια, το οποίο δημιούργησε μια νέα σειρά προβλημάτων. Ο κύριος Τσάχλ Γκέρανς είναι ο εισηγητής μας για το θέμα αυτό. Ε, σε αυτό το στάδιο της ε, συζήτησης θα ακούσουμε τον κύριο Γκέρνη, ο οποίο θέλει να ακούσει τι δικέ σα απόψει, χωρί να έχουμε κάποια έκθεση, κάποιο προσχέδιο έκθεση ακόμα. Κύριε Γκέρνη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, όπω είπατε, αυτό που θέλω είναι να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων για να ξεκινήσω να συντάσω ένα προσχέδιο έκθεση και ένα προσχέδιο ψηφίσματο. Ε, για το θέμα αυτό μπορεί να πει κανεί πολλά, αλλά θα το απλοποιήσω ίσω και υπερβολικά να το υπεραπλώσω. ένα δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια επένδυση η οποία θα δημιουργήσει μετά ε, παραγωγή και αυτό είναι καλό. Όμως μπορεί να είναι παράδεκτο, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα να χρησιμοποιηθεί για να ε, πληρώσουμε τρέχουσες ανάγκες. Στην περίπτωση των ιδιωτών αυτό μπορεί να πρόκειται για ένα καταναλωτικό δάνειο, αλλά το κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και με τα κράτη. Γιατί αυτό το τόκος που είναι το κόστος του δανείου το περνάμε στις επόμενες γενναίες. Και αν μιλάμε για έναν ε, ένα πρόσωπο το οποίο δανείζεται σε, σε, σε προχωρημένη ηλικία, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά του θα αναγκαστούν να πληρώσουν όλου αυτού του τόκους όταν θα βρίσκονται πέστε μέση ηλικία. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πούμε και για ένα κράτο το οποίο ε, έχει υπερδανιστεί. Η προσπάθεια που γίνεται εδώ είναι να ε, πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κάποιους κανόνες τουλάχιστον ε, έτσι ώστε αν όχι να λύσουμε την κρίση χρέου στην παγκόσμια, τουλάχιστον να ε, φροντίσουμε να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι συνέπειε και, και τι ζημίε που προκαλούμε με τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι στους θεσμικούς ε, παράγοντες, στα, στα κράτη και τις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτήν την καταστροφική ε, αυτοτροφοδοτούμενη κρίση που ξεκινάει με μια οικονομική κρίση και μετά οδηγεί σε φτωχοποίηση του πληθυσμού. Ε, Θα προσπαθήσω να δομήσω ότι την, την έκθεση μου σε δύο σκέλη. Το πρώτο θα παρουσιάζει τι λειτουργεί, τι, είναι σωστά καμωμένο και το δεύτερο θα εστιαστεί στα προβλήματα, τι θα έπρεπε να αλλάξει ε, στο επίπεδο το θεσμικό και το, ε, το πολιτικό. Λοιπόν, τι δεν λειτουργεί. Δεν έχουμε συνεκτικές μακροοικονομικές πολιτικές. όταν έχουμε μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα χρέους, ε, δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και πολλές φορές το κοιτάμε με μια μυρολατρεία το πρόβλημα ε, διαφθοράς που μπορεί να υπάρχει. Πολλές φορές ε, ο υπερδανισμός τελικά οδηγεί σε προβλήματα σε εκείνα τα πρόσωπα τα οποία είναι ακριβώς εκείνα που έχουν τη λιγότερη ευθύνη, τη λιγότερη ευθύνη για τον υπερδανισμό της χώρας τους. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για ένα δάνειο από κρατική πηγή είτε από ιδιωτική. Ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες αυτό τις οδηγεί σε περιθωριοποίηση και, τις, ε, και έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν ποτέ να πάρουν στα χέρια τους την, τα μακροοικονομικά τους. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει ε, είναι ότι θα... αυτό, που δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή είναι να αγνοούμε την επίσημη την παραοικονομία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και να, να, να αναγνωρούμε το, τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία και το γεγονός ότι αυτή η κρίση χρέους τους παρεθωριοποιούν ακόμα περισσότερο. Επίσης, ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ότι αυτό το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών, χωρών πολλές φορές χρηματοδοτεί πλέον ε, πολιτικέ πολιτικές ελίτσες αυτές τι μέτρα χρειάζονται. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία να φροντίζουν έτσι ώστε να μην πέσει σε, ένα, ε, σε μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα, ιδιαίτερα μια αναπτυσσόμενη χώρα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη, έχουμε τέτοια παραδείγματα στην Αφρική. Ε, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά που, στα οποία οδήγησε η συμφωνία του Σουάσιγκτον, το τράστι του Σουάσιγκτον. Πολλές φορές ο, ο, δότηση, μάλλον η, η, λήψη δανείων από μια αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί να γίνεται χωρίς μια πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Ε, αυτό αφορά και τους ε, διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και την, ε, τα δάνεια από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να φροντίσουμε το χρέος της χώρας να παραμένει σταθερό, γιατί εάν μια χώρα πάψει να έχει πρόσβαση στι αγορέ για να μπορεί να δανειστεί, αυτό οδηγεί αμέσως και στο θέμα με επενδύσεων αυτήν. Άρα χρειάζεται να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενες χώρε να χειριστούν τα δημόσια οικονομικά του και ιδιαίτερα στους εξή την, την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου την ενίσχυσή τους, στην προσπάθειά τους να θέτουν εκείνη, εκείνα τα κοινοβούλια τι προτεραιότητε του προπολογισμού. Είναι απαραίτητο όταν μια χώρα δεν έχει πια τη δυνατότητα να δανειστεί από τις αγορέ, να, να αναζητήσει άλλες πηγές. Και στην έκθεσή μου θα καταγράψω μια σειρά μέτρων που μπορούν να ληφθούν ε, όταν ένα κράτο βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί να χειριστεί μόνο του. Κάποιες τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να τι προβλέψουμε, αλλά όχι πάντοτε. Δεν ε, δικαιούμαστε να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός της χώρας αυτής εξαιτία του χρέους τη. Θα πρέπει να βρούμε άλλου ε, τρόπους βοήθειας, όχι για να βοηθήσουμε μια τυχόν διεφθαρμένη κυβέρνηση, αλλά για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Ε, Επομένω, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα τι επιπτώσει που θα έχει η δότηση στου ιδιαίτερα στους πιο φτωχού. Και επίσης θα πρέπει να, θέσουμε, ε, να αμφισβητήσουμε τη λογική που λέει ότι η διαγραφή ενός χρέους αποτελεί ε, βοήθεια προ μια χώρα αυτή τη στιγμή ένα κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να ε, αποπληρώσει το χρέος του. Θα πρέπει να ε, αξιολογηθεί κατά πόσον τελικά αυτό το δάνειο είχε βοηθήσει στην ανάπτυξή του. Αν έχουμε ε, τους πολιτικούς ή τη δημόσια δίκηση, η τη δημοσια έχει όντως προσπαθήσει να επιτύχει την ανάπτυξη, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους εκείνοι οι οποίοι δίνουν δάνεια για την ανάπτυξη, για, ως δάνεια αναπτυξιακής βοήθειας. θα, ε, και ε, οι ευθύνε πρέπει να λεφθούν και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του δανειολήπτη και από την πλευρά του Ο στόχος, ο κύριος στόχος λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε απέναντι στις χώρες ε, τις ε, αναπτυσσόμενες είναι πρώτα απ' όλα να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Γιατί η φτώχεια είναι παραβίαση ε, ανθρώπινου δικαιώματος. η αρχή μας είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και να μην καταδικάζουμε ε, τους πολίτες μιας χώρας εξαιτίας μιας πιθανώς ατυχούς διαχείρισης των μακροοικονομικών της μιας χώρας. Ε, ναι, μπορεί να, έχουν, να φέρουν ένα μέρος της ευθύνε οι πολίτες, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες. Σας περιέγραψα κάπως την φιλοσοφία α, της έκθεσης που θα προετοιμάσω. Ε, πρόκειται για μια πολιτική τοποθέτηση απέναντι σε ένα πρόβλημα ε, της ε, και παγκόσμιο. Ε, πολλές φορές αυτά τα ζητήματα δεν συζητούνται ή δεν συζητούνται επαρκώς στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας επειδή δεν θέλουμε να επέμβουμε στα εσωτερικά, λέμε, της χώρας. Όμως, πρέπει ε, να φροντίσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι εταίροι μας στην Αφρική και, και οπουδήποτε αλλού. Ε, αυτή είναι η γενική πρόταση που κάνω προς τους συναδέλφους. Ελπίζω να ε, μπορέσουν να με βοηθήσουν με τις σκέψεις τους αυτή τη συζήτηση τώρα, έτσι ώστε να καταλήξουν σε μια περιστατωμένη έκθεση. Σε ευχαριστώ, Σάρλ. Έχουμε τώρα τους κοιόδους εισηγητές, ο Μπόκταν Βέντα, εκπρόσωπη τον κύριο Σένφελντ, από ό,τι ξέρω. Ναι, ευχαριστώ. Θα μιλήσω πράγματι εκ μέρους ε, του συναδέλφου μου, αλλά στη μητρική μου γλώσσα εγώ. Το χρέος των αναψωμένων χωρών είναι ένα άκρος πολύπλοκο ζήτημα και πολλές φορές έχει συζητηθεί και σε διάφορες ε, διασκέψεις των ΗΕ Εθνών σε σχέση με την ανάπτυξη. Τα δάνεια επιτρέπουν σε πολλές ε, χώρες ε, ουσιαστικά να αυξήσουν τις εσωτερικέ του επενδύσεις. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση. Δεν υπήρχε μετάφραση προς τα γαλλικά. Τώρα υπάρχει. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, είναι το Σάρλ. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Ωραία, Μπόγκταν συνέχισε. Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών είναι άκρος πολύπλοκο και έχει συζητηθεί πολλές φορές ε, και στις διασκέψεις ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Τα δάνεια επιτρέπουν σε πολλές ανυψόμενες χώρες τελικά να αυξήσουν επιτυχώς την κλίμακα των ιστορικών επενδύσεων, αλλά η χρέωση, το χρέος αυτό σε κάποιες χώρες συνιστά ένα μεγάλο άχθος και τους επηρεάζει αρνητικά και στο να κρατήσουν κάποια επίπεδα ανάπτυξη αλλά και στο να ικανοποιήσουν τι βασικέ ανάγκε των πολιτών του. Σε ό,τι αφορά την αφαιρεγκαιότητα άλλων ε, φορέων, εκεί μπορεί ε, να ε, λυθεί το πρόβλημα για τη δικαιοσύνη με την κήρυξη σε πτώχευση. Όταν όμως ένα κράτο είναι χρεωμένο, αυτό έχει πάρα πολύ βαθιές οικονομικέ και κοινωνικέ επιπτώσει. Για δεκαετίες λοιπόν έγιναν συζητήσει και δικαιολογημένα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διεθνούς μηχανισμού διαχείρισης ε, του χρέους ε, χωρών. Σημαντικές διατάξεις για τα θέματα αυτά περιλαμβάνει η Συμφωνία του Μοντερέι του Μαρτίου του 2009. Συμφωνία για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες. Και από ό,τι φαίνεται, το βασικό ε, ζήτημα, ο βασικός παράγοντας για τη διαχείριση του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών είναι το ζήτημα της λογοδοσίας της ευθύνης και των φορέων που δανειοδοτούν τις ανεψόμενες χώρες. Θα πρέπει να προβαίνουν σε μελέτη της φερεγγιότητας του κάστοτε κράτους για να αποφεύγονται μίζωνες κραυδασμοί και ε, σε περίπτωση συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών. Κάτι ακόμη σημαντικό είναι ότι και οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι στη συμπεριφορά τους, γιατί ναι μεν η ακύρωση χρέους μπορεί να βοηθήσει απελευθερώντας πόρους για άλλους στόχους. Αλλά αυτού του είδους η βοήθεια θα πρέπει να συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις προκαταρκτικές, δηλαδή καταπολέμηση διαφθοράς, διαφάνεια δημοσιοοικονομικών, διαφάνεια μεταφορών πιστώσεων, χρηστή διακυβέρνηση. Ο κ. και ο εισηγητής, ε, πιστεύω ότι θα υπάρξει πολύ καλή συνεργασία και με τον εισηγητή και τους άλλους κοιότητες. Αυτά. Ο κ. Βουντζούλικα, το εκμέσιο των Σελίδων Δημοκρατών. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά ε, δέχθηκα την ανάληψη αυτής της έκθεσης. Ε, για ποιο λόγο. Διότι κυρίε και κύριοι όπως γνωρίζετε η δανειοληψία είναι ένα σημαντικό σημείο ε, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μπορεί να βοηθήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως τα υψηλά επίπεδα χρέους είναι ένα βάρο που μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσει αστάθεια και δημιουργήσει σημαντικού κινδύνους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρε χώρες και που έχει οδηγήσει σε μείωση του χρέου και η διεθνή κοινότητα έπαιξε προ αυτό σημαντικό ρόλο, το θέμα τη βιωσιμότητα εξακολουθεί να μα απασχολεί και να μα ανησυχεί. Η παροχή βοήθεια ανεψόμενε χώρε για να έχουν ε, βιώσιμα μακροχρόνια χρέη θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Το ίδιο και η στήριξη και η βελτίωση της δανειλητικής ε, ε, ικανότητας. Όμως εξελίσσεται το τοπίο της δανειοδοσίας, δανειοληψίας και, και τα εργαλεία τα σχετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να αναλύουμε και να έχουμε μία προσέγγιση στραμμένη πιο πολύ προς το μέλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο το πώς μια χώρα υποτίθεται ή κρίνεται ότι έχει βιώσιμο ή μη βιώσιμο χρέος. Η προσέγγιση, για παράδειγμα, των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών βασίζεται σε αναλύσεις οικονομικής ανάπτυξης, εξωτερική εμπορική δυναμική και τους ε, διαθέσιμους πόρους, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα οι άλλες διατάξεις και θα πρέπει αυτή τη βιωσιμότητα να τη δούμε και στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της, ε, του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης το ρυθμιστικό κενό που υπάρχει. Μεγάλο ποσοστό πιστής δεν καλύπτεται από κάποια ρύθμιση. Ένα σημαντικό μήπως τα εμπρός θα ήταν η δημιουργία ένας κοινού γενικού κανονισμού και αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης για οριζόντιες τακτικές αναλύσεις. Αυτή την έννοια η διάσκεψη του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ε, ανάπτυξη έχει σημαντικό ρόλο. Αλλά μπορεί να δυσκολευτεί να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό γιατί δεν έχουν οι χώρες ακόμη στο σύνολό τους ε, ενστερνιστεί τι αρχέ και έχουν βέβαια προσχεθεί το πράξο στο προσεχέ μέλλον. Αυτά λοιπόν για μια ακόμη φορά ευχαριστώ και θα συνεργαστώ στενά όπως πάντοτε με τον Ισίδη και τους άλλους και ό,τι εισηγητές για να πετύχει σημαντική, πολύ σημαντική αυτή έκθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο Τζούτη της Αργεντίνη επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. ο εισηγητής έθεσε κάποιες ερωτήσεις και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύομαι να απαντήσω. Προσπαθώ ακόμα να αντιληφθώ τι ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θα οδηγήσει σε μια ευρία εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουν οι χώρες το χρέος τους και πώς ε, υπερχρεώνονται ή εξετάζουμε ευρωπαϊκές πολιτικές και τον τρόπο με τον οποίο εμείς βοηθούμε ή δεν βοηθούμε τις ε, ε, χώρες υπό ανάπτυξη ε, με το χρέος τους. Δεν είμαι βέβαιη προς τα που θέλετε να κατευθυνθείτε. Ε, εγώ θυμάμαι ότι ε, όταν είχαμε το Ιωβιλέο το 2000, πριν από 17 χρόνια, γινόταν συζήτηση για το χρέος και αφορούσε το ταχθές χρέος. Χρέος σε αναπτυσσόμενες χώρες, που υπήρχε διότι ο δικτάτορας αγόρασε ένα πολύ μεγάλο στόλο αεροπλάνων. Για παράδειγμα δεν μπορούσε να αποπληρώσει, τα αεροπλάνα ποτέ ε, δεν ήταν προς όφελος των πολιτών και αυτό το χθέως ε, ε, το θέμα ήταν ποιος είναι υπεύθυνο για αυτό το χρέος, έπρεπε να πουληθούν τα αεροσκάφη ε, για να αποπληρώσει η χώρα ή ε, τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτή ήταν η συζήτηση. Και η ευθύνη η δική μας ε, είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την εξετάσουμε. Μία από τι νέε πτυχές που έχουν ανακύψει για την ομάδα μου είναι το blending. προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε συνδυασμό με κάποιο ελκυστικό δάνειο. και πρέπει να προσφέρεις λοιπόν βοήθεια, πρέπει να υπάρχει και το δάνειο. Τι σημαίνει ε, αυτό για την αναπτυσσόμενη χώρα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις πολιτικές για τη βοήθεια στο χρέος ε, ε, πριν από 17 ε, χρόνια συζητούσαμε τις ε, εκστρατείες για τους στόχους της χιλιοτίας και το Ιαβιλέο και τότε ήταν συγκεκριμένα τα μέτρα αλλά δεν τα έχουμε πετύχει. Τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τη βιωσιμότητα του χρέου. Δεν επιτυγχάνουμε το 0,7% σε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ε, αλλά ε, βασιζόμασταν και μετρούσαμε στο ποσοστό και την, ε, στην εξυγίανση του χρέους, διότι ακόμα δεν είναι υγιές αυτό το θέμα αυτό. Τώρα, το σημερινό χρέος από πού προέρχεται. Είναι ιδιωτικό δανισμό, διότι φαίνεται να είναι όλο ένα και περισσότερο συχνό. Ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν ενα και περισσοτερο συχνο ιδιωτικοι φορει που παρεχουν ομολογα και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, αγοράζουν αυτά τα ομόλογα ή εμείς ακόμα ε, δανείζουμε και οδηγούμε σε χρεοκοπία τις χώρες αυτές. Πρέπει να το δούμε λοιπόν και το θέμα αυτό. Εμείς ε, πρόσφατα συμφωνήσαμε ως πράσινοι και σε μία νέα πολύ προοδευτική μέθοδο για να προχωρήσουν ε, ε, οι υποδομές σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και πάλι συνοδεύεται από δανεισμό για αυτά ε, τα έργα υποδομών. Δεν τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, εμείς έχουμε και την εσωτερική μας εμπειρία ως Ευρωπαϊκή Ένωση με χρέος που δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Σκεφτείτε την Ελλάδα. Βοηθήσαμε να διασωθούν τράπεζες, τράπεζες οι οποίες ήταν υπερχρεωμένες. είδαμε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να επιτρέπουν ε, να πουληθούν ε, μεγάλες ε, στρατιωτικές υποδομές στην Ελλάδα και να χρεωθεί η χώρα στη Γερμανία. Έχουμε λοιπόν και μία μικρή δυνατότητα να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν χρεώνονται μόνο οι χώρες και δεν είναι υπόλογες μόνο αυτές οι οποίες υπερχρεώθηκαν, αλλά και αυτοί που βοήθησαν να υπερχρεωθούν αυτές οι χώρες. Πρέπει να δούμε τρόπους λοιπόν με τους οποίους ε, μπορούμε εμείς ως Ευρωπαίοι να σταματήσουμε να ζημιώνουμε αυτές τις χώρες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες σαφείς συστάσεις. Ε, είδαμε και συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας και το ε, χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών ήταν υποσυζήτηση, αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε συστάσεις για το πώς Μπορούμε να το εφαρμόσουμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα πράγματα. Αυτέ είναι συστάσει για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώ μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συστάσει. Η Λόλα Σάντσε. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες παγιδεύτηκαν εδώ και δεκαετίες με πολλέ απώλειε, συνεχιζόμενε απώλειε. Ε, δεν ήταν επαρκώς ε, ε επαρκής μάλλον συγγνώμη, χρηματοδότηση και δεν μπορούσαμε να καλύψουμε το χρηματοδοτικό χάσμα. Τελικά βρίσκονται σε ένα αένα χρέο αυτές οι χώρες και αυτό το νιώθουμε και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση η οποία χτύπησε διεθνώς και είδαμε πάρα πολλές ε, ε, χρηματοδοτήσεις από το δημόσιο κορβανά για αποτυχημένες τράπεζες και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν σε διεθνές επίπεδο και στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και οι βιομηχανοποιημένες χώρες αντιμετώπισαν αύξηση στο επίπεδο του χρέους. Το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη έφτασε σε ε, ύψη τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ σε καιρό ειρήνης. Το χρέος όμως σε χώρες ε, αναπτυσσόμενες ε, όπου υπάρχουν και ανάγκες χρηματοδότησης λόγω της μείωσης της ενίσχυσης και των προβλήματα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για σύμπτωμα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και της αυξημένης φτώχειας. Το χρέος αρκετών χωρών δεν είναι απλώς μη βιώσιμο, αλλά πολύ μεγάλο τμήμα των δημόσιων χρεών προκύπτει και από υπερχρέωση ε, και πολύ σημαντικές συνέπειες για το κλίμα ή προέκυψαν λόγω αγοράς ε, ε, εξοπλισμού, οπλικών συστημάτων ή και όπλων. Οι δανειοδότες ε, κυριαρχούν γιατί είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες ε, οι οποίοι διέπουν τα παιχνίδια του χρέους τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθορίζουν τους κανόνες που καθορίζουν κατά πόσον μια φτωχή χώρα μπορεί να αποπληρώσει ή μη το χρέος της. Πρόκειται για το πλαίσιο βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό το πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη του στις ανθρώπινες ανάγκες και βασίζει τι αναλύσεις του σε πολύ συγκεκριμένε περιορισμένες ε, ε, συνιστώσεις και φυσικά διονύζεται η φτώχεια και δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Και οι είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες για την επίλυση της κρίσης. Αντίθετα με τις επιχειρήσεις ή τους ανθρώπους δεν υπάρχει ένα σύστημα για τις χώρες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος τους και δεν υπάρχουν και μηχανισμοί που επιτρέπουν οι δανειοδότες ε, να λογοδοτούν για τα επισφαλή δάνεια τα οποία οδηγούν τελικά σε ε, παράνομο χρέος. Στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες ε, αναδιάρθρωσης στον τομέα αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικά μπλοκ τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί. Ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα για το κυρίαρχο χρέο απαιτεί κατά την άποψή μα ένα διεθνή μηχανισμό που θα λαμβάνει υπόψη του ε, διεθνεί πόρου που πρέπει να έχει μια χώρα για να μπορέσει να αποπληρώσει τι υποχρεώσει τη και να μπορέσει να καλύψει και τι κατάλληλε υπηρεσίε για του πολίτε. Χρειαζόμαστε κάτι λοιπόν που θα βασίζεται στι ανθρώπινε ε, ανάγκε για τη βιωσιμότητα του χρέου. Να είναι εξάρτητο από του πιστωτέ και του δανειστέ ε, και φυσικά να ε, ε, βρίσκεται σε ένα ε, ανεξάρτητο βήμα, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Έθνη ή τα ανεξάρτητα δικαστήρια. Πρέπει να περιλαμβάνει πολυμερή διάσταση και να καλύπτει όλες τις ανάγκες των χρεών πολύ γρήγορα και να καλύπτει όλες τις χώρες που μπορεί να κινδυνεύουν να βρεθούν υποχρεωμένε. Και φυσικά πρέπει να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα να εισακουστεί κανεί και να παρουσιάζονται και να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία. Εάν μια χώρα θεωρεί ότι έχει βιώσιμο ή μη βιώσιμο ε, χρέος, ε, ε, το τι κάνει η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο και πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η διεθνής πιστοτική κοινότητα. Πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες εξωτερικού εμπορίου και διαθεσιμότητα εξωτερικών πόρων και αν μπορεί μια χρεωμένη χώρα να αποπληρώσει ή μη το χρέος της και να τηρήσει τις υποχρεώσεις δεν λέγονται πάρα πολύ για τι συνέπειε για την ανθρώπινη ανάπτυξη στο θέμα αυτό. Η έννοια της βιωσιμότητα του χρέου πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και του σπόρους που χρειάζεται οι αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορέσουν να καλύψουν την ένδια και την ανισότητα και φυσικά να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και γι' αυτά πρέπει να γίνεται ανάλυση του χρέου και λαμβάνοντα υπόψη μια ανθρώπινη συνιστόσα πρέπει να λαμβάνουμε και τον άνθρωπο υπόψη για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του χρέους. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρενς για την παρέμβασή του, διότι και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή κοινή βάση για να συνεργαστούμε στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ζήτησα ήδη συγγνώμη από τον εισηγητή, γιατί δυστυχώ θα πρέπει να φύγω. Έχω μια άλλη συνάντηση και δεν θα μπορέσω να ακούσω την απάντηση που θα, σας, που θα μου δώσει. Όμως, εγώ θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Τι γίνεται όταν έχουμε μια χώρα η οποία έχει επωφεληθεί από μια διαγραφή του χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα ή από κάποιο διεθνή οργανισμό και μετά από λίγα χρόνια βρίσκεται πάλι υπερχρεωμένη εναντί κάποιου, κάποιου άλλου πιστωτή της Κίνας ή οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό ως πρόβλημα, ως θέμα, ως ενδεχόμενο για να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα. Η Πρόεδρος, ε, έχουμε τον κύριο Κόβατ από από τη Γενική Διευθυνσή Αναπτυξιακή Συνεργασία. Δεν γνωρίζω αν έχει αναλάβει κάποια σχετική πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν αναφέρετε το θέμα αυτό όταν έχετε διτημερεί επαφέ για αναπτυξιακή συνεργασία, χρήσιμο θα ήταν να μα ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Βεβαίως, πολλά από τα θέματα που ακούστηκαν στη συζήτηση είναι ε, ζητήματα ενδιαφέροντος ή και ανησυχία και προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε την βιωσιμότητα των διαφόρων προγραμμάτων ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες εκ των προτέρων. Βλέπω ότι αλλάζει κάπως η δημόσιος διάλογος για πολλές δεκαετίες, για τα τελευταία 15 χρόνια υπήρξαν εξτρατείες κατά της υπερχρέωσης των αναπτυσσόμενων κρατών, οι οποίες πράγματι είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά το χρέος τους ε, μέχρι το 2010-2011, όμως έχει αντιστραφεί αυτή η πορεία και έχει ξαναρχίσει το χρέος των αναπτυσσόμενων κρατών να αυξάνεται από τότε και μετά. Αν κανείς αναλύσει τη δομή του χρέους, θα διαπιστώσει ότι στην υποσαχάρια Αφρική ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 18 ποσοστίες μονάδες, που είναι πολύ σημαντικό. Ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνεισφέρουν σε αυτό. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν σημαντικές ανάγκες ανάπτυξης. Και αυτό το αναγνωρίζουμε και στο θεματολόγιο μας για την ανάπτυξη, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες επενδύσεις στις χώρες της Αφρικής και δημόσιες και ιδιωτικές. Αν αυτές οι επενδύσεις αξιοποιηθούν με τρόπο παραγωγικό, μπορεί να φροντίσει κανείς να διαχειρίζεται το χρέος του αποτελεσματικά. Όμως γνωρίζουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση του χρέους ε, των αναπτυσσόμενων χωρών είναι το γεγονό ότι τα επιτόκια διεθνώς είναι πάρα πολύ χαμηλά και αυτό οδηγεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ακολουθούν πολιτικές για να μεγιστοποιήσουν τα δικά τους κέρδη με αποτέλεσμα να ε, ψάχνουν για όλο περισσότερο ε, μεγαλύτερη δανειοδότηση και αυτό οδηγεί σε έκδοση όλο και περισσότερο ομολόγων από τις αναπτυσσόμενες χώρες και βρίσκουν ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι χώρες αυτές, στην Ευρώπη ή αλλού. Η διεθνή κοινότητα με το θεματολόγιο της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, Financing for Development, του 2015, έχει αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να αυξηθούν οι επενδύσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα δισεκατομμύρια πρέπει να γίνουν 3 εκατομμύρια και αναγνωρίζει ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα αποτέλεσμα και στο επίπεδο του χρέου, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μια εκ των προτέρων στρατηγική διαχείρισή του. Η Επιτροπή συνεργάζεται με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα για τα θέματα αυτά, γιατί είναι οι δύο οργανισμοί, οι θεσμικοί οργανισμοί που ασχολούνται με τα ζητήματα ε, του χρέου σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, έχει ήδη αναφερθεί ότι υπάρχει το πλαίσιο για τη βιωσιμότητα του χρέους του Διεθνούς Νομικοσματικού Ταμείου, το οποίο εφαρμόζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες και το οποίο πρόσφατα επικοινοποιήθηκε. Η ε, Παγκόσμια Τράπεζα έχει επίσης ένα ταμείο για τις υπερχρεωμένες χώρες στην οποία ε, και, ε, συνεργαζόμαστε με μεμονωμένες αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουμε να αξιολογήσουν τον κίνδυνο ε, εξαιτία του χρέους, τον κίνδυνο εξαιτία των νομισματικών διακυμάνσεων ε, ή οποιοδήποτε άλλη μορφή κίνδυνου. Υπάρχουν επίσης κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, των στατιστικών στοιχείων. Ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί σοβαρά. Σε πολλές χώρες υπάρχει κρυμμένο, κρυφό χρέος. Ε, το οποίο έχει προέλθει από κάποια δάνεια τα οποία ίσως να μην έχουν καταγραφεί στα δημόσια οικονομικα ή από κάποια δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί από συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Και αυτό το, ε, το, το χρέος μπορεί να παραμένει κρυφό ακόμα και από τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν έχουν ε, χώρες αυτές ένα σύστημα δημόσιων λογιστικών το οποίο θα επέτρεπε στο Εθνικό Κοινοβούλιο να ασκήσει τις ελεκτικές του αρμοδιότητες και να γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο του χρέους. Αυτό δημιουργεί προβλήματα που βγαίνουν και μεγενθύνονται με την πάραδο του χρόνου. Μιλώντας τώρα για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε σχέση με μεμονωμένες τώρα χώρες, προσπαθούμε πάντα να έχουμε έναν πολιτικό διάλογο με τις αρχές των χωρών αυτών η κατάσταση με το χρέος μιας χώρας πρέπει να τη βλέπει πάντα κάνει σε συνάρτηση με τη γενικότερη ε, μακροοικονομική της πολιτική και την, τα δημοσιονομικά της. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν πολλούς φυσικούς πόρους στη διάθεσή τους ε, και άλλες χώρες οι οποίε έχουν καταφέρει να έχουν πιο περισσότερο διαφοροποιημένε οικονομίε. Οι χώρε εκείνε οι οποίε έχουν τα πιο άμεσα και σοβαρά προβλήματα διαχείριση χρέου είναι εκείνε οι οποίε παραδοσιακά εξάγουν πετρέλαιο, μεγάλε ποσότητε πετρελαίου, γιατί εξαρτούνται από τι διακοιμάσει στην τιμή του πετρελαίου ή άλλων φυσικών πόρων. Ε, κατά τα άλλα, βέβαια, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μετά από χώρα σε χώρα. Ε, εκείνες οι οποίες ε, χώρες καταφέρνουν να εξάγουν μια ευρία κάμα, ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, καταφέρνουν να ε, κρατούν το έλλειμμά τους χαμηλό και άρα να διαχειρίζονται καλύτερα και το χρέο τους. Αυτά κατά βάση κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι ακόμα ενδιαφέρον, το οποίο δεν ανέφερα, είναι το εξής Συμφωνούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί και αυτή για το γεγονό ότι δεν υπάρχει ένα διεθνέ πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του χρέου. Το οποίο σημαίνει ότι όταν φτάνει σε μια ε, κατάσταση ε, μια χώρα να μην μπορεί να ε, αναχρηματοδοτήσει το, το τη, γίνεται μια διαδικασία ad hoc και πάντοτε υπάρχει ένας, ο κίνδυνο να υπάρξει ένα σημαντικό αριθμό πιστωτών που δεν έχουν διάθεση να συνεργαστούν με αυτή την αναδιάρθρωση, να, να μπουν στην αναδιάρθρωση. Ε, εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση μας. Γιατί πηγαίνουμε όλο και περισσότερο προς ιδιωτικούς πιστωτές, όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο ε, κρατικούς πιστωτές από ότι στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε το το λεγόμενο κλαμπ των Παρισίων, χώρες ευρωπαϊκές, τις Ηνωμένε Πολιτείε και μεγάλες αναπτυγμένες χώρες που δάνειζαν κατά κύριο λόγο. Τώρα έχουμε όλο και περισσότερο ε, διεθνή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ακόμα και ε, τις ε, αναδιόμενες οικονομίες. Και αυτό αλλάζει την κατάσταση. Τώρα όσον αφορά την τη χρηστή διαχείριση όσον αφορά τον δανεισμό. Υπάρχουν κατευθυντήριε οδηγίες του ΟΗΕ, ένα κατάλογο κατάλογος αρχών που και οι πιστωτέ και οι δανειστέ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη του. Αλλά φυσικά είναι ε, ένα καλό έτσι ε, έγγραφο το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Το ζήτημα έχει επίση συζητηθεί στο πλαίσιο των G20 και κατέληξαν σε ένα κείμενο συμπερασμάτων πέντε σελίδων. Και πάλι ε, ένα, μια κατάλογος αρχών που κάθε πιστωτής και κάθε δανειζόμενος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του. Αλλά και πάλι ε, αυτά, αυτές οι αρχές μένουν στα χαρτιά θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται και αν εφαρμόζονται. Αυτά από την πλευρά μας, αυτές τις πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις, όπως έλεγα, και ε, σε συστηματική ε, βάση τα χρονικά διαστήματα ε, ενημερώνουμε για τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Σάρλ, για τη δευτερολογία του. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, στο ερώτημα της κυρίας Αργεντίνη. Νομίζω ότι είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση ότι η, σχέση για το, η έκθεση για το σχέση στόχο έχει να βάλει όλους τους φορείς αναπροσανευθυνών τους, δηλαδή τους πιστωτές, ιδιωτικούς και δημόσιους. Και τους ε, οφειλέτες όμως. Πώς θα φερθούν ένα από των ευθυνών τους. Ε? Εγώ σκέφτηκα ένα κώδικα συμπεριφοράς. Υπάρχουν κανόνες, αν δεν είναι κωδικοποιημένοι, το είπε και η Κομισιόν. Άρα θα έπρεπε ίσως να δούμε πώς μπορούμε να καταστήσουν πιο υπεύθυνου ε, όλους αυτούς τους ε, φόρους. Και πρώτα απ' όλα, εγώ στο επίκεντρο θέλω να βάλω την ευρωπαϊκή απάντηση. Και η ευρωπαϊκή απάντηση είναι ένα ερώτημα. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε το χρέος. Είπατε ότι δεν πρέπει να δανείζουμε ελαφρά την καρδία και θα πρέπει να αποτρέπουμε τους ε, φορείς παρεμβαίνουν. δυτικοί πιστωτέ. Ποια είναι η ευθύνη των κρατών μελών και τη Ένωση. Αυτοί δεν δανείζουν ελαφρά την καρδία. Κατά το παρελθόν το έκαναν γιατί θα τους έσωζαν, θα τους έσωζαν. Και επειδή βλέπαμε ότι επίκειτο μια μεγάλη κρίση, το είδαμε το 2007 κρύφτηκαν πίσω από την αρχή του big to fail οι ιδιωτές πιστωτές και μετά βέβαια λήφθησαν μέτρα για να τους ε, καταστήσουν πλέον υπεύθυνου για την συμπεριφορά τους. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να απαιτήσουμε μια τράπεζα να δίνει δάνειο σε έναν που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι και πρέπει να έχει ένα αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης πολύ σημαντικό για να μειώσει το κίνδυνο της τράπεζας, το ρίσκο της τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Αν το κάνουμε αυτό, γιατί να μην υιοθετήσουμε την ίδια προσέγγιση και όταν θέλουμε να δώσουμε δάνειο σε μια αναπτυσσόμενη χώρα ή σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Έχουν και αυτή την ευθύνη τους και πρέπει σε αυτή την οδό να επιμείνουμε. και τους θεσμικούς πιστωτές Παγκόσμια Τράπεζα και Δέλτα Νιτάφ. Επίσης και αυτούς πρέπει να τους κάνουν πιο υπεύθυνους. Το Δέλτα Νιτάφ δίνει πολύ βράχη πρόθεσμα δάνεια που πρέπει μέσα σε σύντομη περίοδο τριών ετών να έχουν ε, εξυπηρετηθεί. Η Παγκόσμια Τράπεζα πιο μακροπρόθεσμα δάνεια. Και ιδίω σε αυτή την εποχή δεν ήταν πάντα έτσι. Ένα μέρος της λύσης είναι, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας, αν ένα κράτος δεν μπορεί να τα καταφέρει, να αποπληρώσει, δεν πρέπει να δανειστεί. Δεν του δίνουμε άλλα δάνεια. Αν έχει καταστραφεί μια χώρα και επειδή κατατρίχεται από τη διαφθορά και μετά πλέον καταραίει, καταστρέφεται γιατί έχει κάνει μεταστάσεις σε όλον τον δημόσιο ιστό αυτή η διαφθορά, όπως και στον οικονομικό ιστό της χώρας, σημαίνει ότι πρέπει να θεραπευτεί το πρόβλημα και πρέπει να επιβάλλονται όροι και προϋποθέσεις από την εταιρική σχέση, να αναζητούνται χώροι για την κοινωνία των πολιτών, που να μπορέσει να παρέμβει και που δεν μπορεί το κράτος να παρέμβει. Σημαντικό είναι λοιπόν, αντίστοιχα, να έχουμε και αρκετά μέσα στη διάθεσή μας, για την χρηματοδότηση προγραμμάτων, σχεδίων ή να παρέχουμε μια δημοσιονομική στήριξη. Πάντα υπάρχει μια ένας διάβολος που θα δουλέψει καλύτερα από κάποιον άλλο. Άρα προσπαθήσουμε να απομονώσουμε ε, κάποιες ε, για να μην επιμολυνθούν από τη διαφθορά εφόσον αυτή ε, κυριαρχεί στη χώρα που θέλουμε να στηρίξουμε και μέσα γι' αυτό υπάρχουν Είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Πρέπει να δούμε την αλληλεπίδραση όλων των μεγεθών που οδηγούν στην επιδείνωση της κατάστασης σε μια χώρα. Και εξωθεί στα ύψη το χρέος. Και ένας παρόντας είναι και η απουσία του κράτους σε σημαντικούς τομείς. Μπορούμε λοιπόν να δράσουμε απέναντι σε αυτούς τους παράγοντες. Εγώ είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Και λέμε και ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πώ θα του κάνουμε πιο υπεύθυνου, πώ θα βάλουμε, φέρουμε ενώπιον των ευθυνών του τους, ε, ε, πιστωτέ. Ένα υπουργό από μια Αφρικανική χώρα ξέφρασε την αγανάκτησή του για την έλλειψη προγραμμάτων ε, καταπολέμηση διαφθορά στη χώρα του. Και για πάνω από μια ώρα συζητήσαμε τι μπορεί να γίνει. Και τελικά καταλήξαμε στο ότι υπάρχουν λίγοι ούτε μία εκατοστή άνθρωποι που σε κάποια χώρα μπορεί να ελέγχουν ε, θέσεις κλειδιά. Και αν αυτοί είναι άσπηλοι και δεν εκτίθενται στη διαφθόρα, μπορούμε να έχουμε μια πρόοδο, αλλιώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και οι χώρες αυτές είναι χαμένες. Ούτε η διαγραφή του χρέους είναι πανάκια. Αυτό που θα μπορούσε να βγάλει τις χώρες από την εξαθλίωση θα ήταν μια προσπάθεια να βελτιωθεί η διακυβέρνηση. Και αυτό ξεκινάει από κάποιες θέσεις κλειδιά που πρέπει να μην ε, επιτρέπουν να υπάρχει διαφθορά και από την ε, ευθυνοποίηση της κυβέρνησης και οι πιο πολλοί δεν έχουν να πούν ε, τίποτα και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και ένας τέος απορφός μου είπε ότι η μόνη συζήτηση που τους ενδιαφέρει είναι η βελτίωση ε, του κλιματισμού της ολομέλειας. Ε, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο. Αυτή την αδράνεια και την κόποση την νοητική των βουλευτών. Μπορούμε να προτείνουμε ανταλλαγές από αυτούς, ε, σε αυτούς τους βουλευτές να έρθουν εδώ, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, στην Επιτροπή Προπολογισμών και να τους μάθουμε τη δουλειά, το επάγγελμα του πολιτικού, του ε, επόπτη, του ελεγκτή. Δεν φεύγουμε άδεια χέρια, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή όταν εδώ και δεκαετίες κάνουμε τις ίδιες διαπιστώσεις. Και είναι αργή η πρόοδος και είναι κουραστικό να επαναρχόμαστε στα ίδια θέματα. Πρέπει να αποθαρρύνουμε Αυτος που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Είναι και εδώ, όχι μόνο, αλλά είναι και εκεί, στις αναψόμενες χώρες. Η κρίση η πολλαπλή και ιδίω η νομισματική, η χρηματοπιστωτική, η δημοσιονομική, η οικονομική, αυτές οι κρίσεις που αλληλεπικαλύπτονταν και που δημιούργησαν μια πολλαπλή κρίση, για να αντιμετωπιστούν πρέπει να σπάσει ο φαύλος κύκλος και να γίνει ένα άρετος κύκλος. Αυτός είναι ο στόχος της παρέμβασής μου, κυρία Σαρτζεντίνη, να φέρω ενώπιον των ευθυνών σε όλους τους φορείς που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση των δημοσίων οικονομικών σε μια χώρα και ιδίω του χρέου, που δεν είναι ένα από πολλά άλλα συστατικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ καλά κάνει η Κομισιόν και υπογραμμίζει ότι υπήρξαν βελτιώσει στο παρελθόν. Θα μπορούσα να κάνω ένα μακρό σκελέστατο επίλογο για όλες τις τεχνικές που κάνουν ένα κράτος να μην είναι κράτος. Αλλά εγώ θα έλεγα η πρόληψη είναι το πάνω. Έχουμε τη λέξη των Παρισίων, έχουμε τις συζητήσει ε, στο πλαίσιο των διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών. Το σημαντικό όμω είναι πολιτική υπεύθυνοι να δείξουν και λίγη φαντασία και δημιουργικότητα. ώστε το χρέος αυτό να ελεγχθεί ή να μειωθεί. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το χρέο. Αλλά και τις μελλοντικέ επιχειρήσεις του Ταμείου Επενδύσεων στην Αφρική. Σε σχέση με αυτό που μας είπε και χθε ο εκπρόσωπο της Κομισιόν για τη χορήγηση εγγυήσεων για τις επενδύσεις. Πρέπει να γίνει εξολόγηση του ρίσκου. Αν είναι λογικός, ο εύλογο, ο εύλογο ο κύριο τότε μπορεί να γίνει μια επιχείρηση, μια ανεπροβλέψιμος. Αν μας δουλέψουν, θα πρέπει να τι σταματήσουμε τι επιχείρησει αυτές όμως. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Βέντα, που νομίζω αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Πενθυμίσει μου λέει του Μόντερεϊ, διαφάνεια, φερεγγιότητα μιας χώρας και αν κατάλαβα, είπε και αυτός ότι η διαγραφή του χρέους δεν είναι πανάκια. Δείχνει μια αποτυχία. Ο κ. Φουντζουλίτσα λέει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα του χρέους, να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και η Αργεντίνη απάντησα. Και ω προς τον κύριο Κορνίγη ήταν ακόμα πιο πολύπλοκο για τους διάφορους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Εδώ υπάρχει μια αλληλεπίδραση και υπάρχει μια αντίληψη ότι μας κοροϊδεψαν. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Κομισιόν που είναι εδώ. Μια γρήγορη, ευσύνοπτη ε, θα είναι η έκθεση για να δούμε ακριβώς τι πολιτικά μέσα μπορούμε να τονίσουμε και να προβάλλουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και να δράσουμε προληπτικά ώστε να ελέγξουμε καλύτερα τα δημόσια οικονομικά χάρη στην χορήγηση υπεύθυνων δανείων και για τους χρηματοδότες, για την ηθική τους, θα θέλω να πω κάτι τελευταίο. Βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται με την παραοικονομία. Αν δούμε πού είναι τα λιγότερα προβλήματα, σε ό,τι αφορά την αποπληρώμη του χρέους, είναι στην παραοικονομία, στην άτυπη οικονομία. Οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις. Και κάτω από τον, πάνω από το 95% ε, που πληρώνονται τα δάνεια αυτά. Και οι οργανισμοί πηγαίνουν και χρηματοδοτούνται στις διεθνείς αγορές και πληρώνουν, ε, παίρνουν πολύ λίγα ποσά, αλλά πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλα επιτόκια. Απαγορευτικά σχεδόν θα έλεγα. Γιατί ο δανειοδότης θα πρέπει να φροντίζει αυτούς που δανείζει να τους πλαισιώνει με συμβούλους που θα τους δίνουν ε, καθοδήγηση για το πόσο θα χρησιμοποιήσουν τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που έχουν πάρει. Μια γυναίκα που δεν είναι καν μορφωμένη μπορεί να τα καταφέρει τόσο καλά γιατί οι άνθρωποι που έχουν μόρφωση δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο για τις υποθέσεις που αφορούν τη χώρα τους. Μακάρι να μπορέσουν όλες οι χώρες να κάνουν τα πάντα για να δείτε τι συνέβησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Λοιπόν, Σάρλ, μπορούμε να περιμένουμε σύντομα την έκθεσή σου. Θα την έχετε σύντομα στην Επιτροπή Γνέφη Καταφατικά. Και λάβατε τα μηνύματα να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες σαφείς συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 13, το πολύ σημαντικό θέμα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο Παουλ Ρούμπιχ. Ε, ε, η γνωμοδότηση είναι για την Επιτροπή Προϋπολογισμών για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίσει ε, τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Ελάχιστα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο σημαντικά στην Επιτροπή μας από αυτή τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά θα ακολουθήσει και η συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πάουλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο είναι κάπως αβέβαιο σε κάποιο βαθμό με τη συνδίκη της Λισαβόνας προβλέπονται τα ποσά και τα τελευταία χρόνια η των κυβερνήσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μειώνουν συνέχεια αυτά τα ποσά ε, που ήταν ε, πάνω από το 1%, 1,4% και τώρα το κατεβάζουν στο 1%. Και λέμε για το 1,24% τώρα. Αυτός είναι ο στόχος, ε, αλλά για την αναπτυξιακή λέμε 0,7% του ΑΕΠ. όχι καθαρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο βέβαια, ούτε μόνο με τις εθνικές πληρωμές. Για κάποιες χώρες μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο πιο εύκολα, κάποιες άλλες χώρες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να καταβάλουν αυτό το ποσό. Υπάρχουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2018 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ανέβει 60 δις 144 δί συνολικά. Και νομίζω ότι το επόμενο πλαίσιο θα πρέπει να δούμε και τη διάρκεια που θα έχει και να λάβουμε υπόψη ε, και τι θα γίνει με τους Βρετανούς, αν θα ε, λάβουμε υπόψη τη δική τους ε, συνεισφορά και τι, πώς θα τα υπολογίσουμε, αν θα είναι 7 χρόνια το επόμενο πλαίσιο, αν θα είναι 5 συν 5. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ακόμη. Για την κατηγορία παριθμών 4 είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε να τηρήσουμε τους διεθνούς μας στόχους, δηλαδή ε, την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτή, αυτός ο στόχος. 2, ε, και 7 είναι πάρα πολύ σημαντικοί στόχοι, ιδίως ε, για τα ταμεία τα οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υγεία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, νέες ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, και απόδοση κτλ. Πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο καλό και για όλες αυτές τις πολιτικές. Και θα πρέπει να δούμε και να προβλέψουμε τα σχετικά κονδύλια στο νομικό πλαίσιο. Επίση, ο ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, θα πρέπει να κινητοποιηθεί να κινητοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, μαζί και με τις λιγότερα αναπτυγμένες χώρες, όπου έχουμε ένα μοντέλο blending και συμπράξεων δημοσιοδιωτικού τομέα που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Νομίζω ότι και για την πολιτική γειτονία είναι κάτι πολύ σημαντικό να ακολουθεί η προσέγγιση του more for more. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον θα χρειαστεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η αναπτυξιακή πολιτική να ληφθεί περισσότερο στο υπόψη, να είναι στο επίκεντρο περισσότερο και στους διακυβερνητικούς ε, τομείς ε, που μέχρι στιγμής δεν είναι υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Επιτροπής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Αν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε και αυτά σε αυτό το προπολογισμό. Νομίζω αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και γιατί θα επηρεαστεί η δημόσια αλλά και κοινή γνώμη, αλλά και γιατί θα είναι πιο αποτελεσματικά τα προγράμματα και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε. Τι άλλους πόρους θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, είτε εθνικούς είτε διεθνείς. Πρέπει πολλά να σκεφτούμε ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε και τα διάφορα καταπιστεύματα που έχουμε δημιουργήσει το μέσο διευκόλυνση για την Τουρκία και πολλά άλλα ζητήματα υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Και αυτό που θέλω τώρα στην προκειμένη περίπτωση είναι να ακούσω την άποψη των συναδέλφων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποια είναι τα βασικά σημεία. Θε συμφωνείτε με αυτά που έχω αναφέρει. και ελπίζω βέβαια ότι ό,τι προτείνουμε μετά θα συζητηθεί και θα ληφθεί υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Εγώ ευχαριστώ. Η Έλλη Λάιν για τους σοσιαλιστές έχει πρώτα το λόγο, σκιώδης συντάκτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρούμπιχ Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας ε, να ετοιμάσει μια αρκετά στεναρή ε, γνωμοδότηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συζήτηση για τον προπολογισμό που δυστυχώς ε, παρουσιάζει μια πολύ ζωφερή ε, εικόνα για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλήσιο. Έχουμε περικοπές στην ανθρωπιστική ε, βοήθεια και επικεντρωνόμαστε μόνο στην άμεση γειτονία και στην ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κοιτάει την ευρύτερη εικόνα. Η νεολαία της ευρωπαϊκής θα είναι δεκαπλάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 και ε, πρέπει να επενδύσουμε σε μακροπρόθεσμους στόχους, γιατί έτσι επενδύουμε και στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξο λοιπόν πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, βάσει και των βιώσιμων στόχων ε, ανάπτυξης που συζητούσαμε σήμερα το πρωί με τους βουλευτές από το Εθνικά Κοινοβούλιο και πρέπει να ενισχύσουμε τις δεσμεύσεις του 0,7. Πρέπει να αναθεωρήσουμε το ανώτατο όριο προς τα πάνω. Θα πρέπει να έχουμε νέους πόρους, συνεπείς, διάφανους και προβλέψιμους τρόπους χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θέτουν η ένδια ενισότητα και η κλιματική αλλαγή. Είναι θέμα συνέπειας και σεβασμού των διεθνών μας δεσμεύσεων. Θα πρέπει να διατηρήσουμε ξεχωριστά την ε, ανάπτυξη και την ε, ε, συνεργασία για την ανάπτυξη από τα άλλα ανθρωπιστικά προγράμματα. Μπορεί να βοηθήσουν φυσικά τα προγράμματα αυτά, δεν το αμφισβητούμε, αλλά δεν είναι κατάλληλη η χρήση ε, των πόρων για την ανάπτυξη. Ε, πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλες παρεμβάσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια. Και ε, ο τίτλος 3 και 4 ε, δεν ε, συζητάται πλέον. Πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχει συνεργασία για την ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τα εσωτερικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα τη μετανάστευση. Το καταπίστευμα για την Αφρική τελικά φαίνεται ότι είναι απλώς για να σταματήσει τους μετανάστες και να σταματήσει τις ροές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει εφταγράμμιση με τις προτεραιότητε των χωρών που δέχονται τη χρηματοδότηση. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ακαιρεότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ε, αναπτυξιακής βοήθειας ε, με κατάλληλη χρηματοδότηση. Η κύρια ε, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να υποστηρίξουμε τις αναπτυσσόμενε χώρε και να μην βασιζόμαστε μόνο στη μετανάστευση και στην ασφάλεια. Και πρέπει επίση να σκεφτούμε και τη το EDF ε, που είναι εξαίρεση για την αρχή της ενότητας του προπολογισμού και ίσως δεν είναι πλέον αιτιολογημένο. Αντιμετωπίζουμε πολλά γνωστά στοιχεία, για παράδειγμα το μέλλον του κοτονού, τις συνέπειες του Brexit ε, και το θέμα των ανωτάτων ορίων, αλλά πραγματικά θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι γενικότερα η απλούστευση των εξωτερικών μέσων είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη συνοχή και να διευκολύνουμε το δημοκρατικό έλεγχο και ε, τα μέσα εκτός προπολογισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για περιορισμένη χρονική διάρκεια και συγκεκριμένους στόχους. Η χρήση καταπιστευμάτων για την περίπτωση, για παράδειγμα, του Ταμείου του Μπακού ή ε, για τους ε, Σύρους είναι κατανοητά, αλλά η καταπολέμηση της ένδυας και της ανεργίας στην Αφρική και ε, τα αίτια της μετανάστευσης δεν μπορεί να είναι ένα κατεπήγον περιστατικό που πρέπει να επιληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να αποτελούν εξαίρεση. Οι νέε δεσμεύσει απαιτούν νέου πόρου, η ανάγκη για καταπιστεύματα για να μπορέσουμε να έχουμε μόχλευση και να αντλήσουμε χρήματα από άλλε πηγέ. Σίγουρα επισημαίνει ότι είναι ανεπαρκή η ευρωπαϊκή πόρη για να επιτύχουμε του στόχου μα και να, δεσμευτούμε τις, ε, ε και να σεβαστούμε Το blending θα πρέπει να συνοδεύεται με διαφάνεια και πρότυπα λογοδοσία. και πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε δεσμεύσει στην αναπτυξιακή συνεργασία και την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά με μια προσεκτική προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες κοινωνικές ε, δικλείδες ασφαλείας, καθώς και δικλείδες ασφαλείας για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επικεντρωθούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής ανάπτυξης, αλλά βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των ανθρώπων. Θα έχουμε ε, τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία με τον κύριο Ρούμπι και τους κοιόδης συγητέ. Thank you very much. Uh, Charles Gerens for the Liberal Group. ευχαριστώ κύριος Γκέρενς. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Ρούπικ για το εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο συντάσσει αυτή την έκθεση. Ουσήθηστε. Η Επιτροπή είναι υπέρ της αύξησης των διαθέσιμων πόρων τους επόμενους το, για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε αυτό είναι 7 χρόνια είτε κάποια άλλη διάρκεια. Και το κοινοβούλιο φυσικά το επιθυμεί αυτό. Ποιο διαφωνεί, ποιο δεν το θέλει, τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, δηλαδή εκείνο που πληρώνει, <laughs> εκείνοι που πρέπει να δώσουν τα χρήματα που πρέπει να βάλουν το χέρι στη ζέπη. Και που πρέπει να βρεθούν από την πλευρά του εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση. Εδώ είναι ο αδύναμος γρήκος όταν πρόκειται να αντιταχθούν στις, ε, στα αιτήματα του Κοινοβουλίου, καταφέρνουν και είναι ενωμένοι και πολύ αποτελεσματικοί, τα κρατημέλη ενώ. Έχουμε δύο σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτα απ' όλα το Brexit. Ε, γνωρίζουμε ότι, ότι από το 2019 θα χάσουμε μια από τις χώρες που ήταν βασικός σημαντικός χρηματοδότης και ε, από τις χώρες που είχαν καθαρή συνεισφορά ήταν μία από τις σημαντικότερες. Αυτό έχει επιπτώσεις γενικότερα για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα για την αναπτυξιακή συνεργασία και αυτή τη στιγμή ε, το, το, το, τα, οι, πόροι οι οποίοι δίνει η Βρετανία δεν ε, θα πρέπει να, να καλυφθούν από κάπου. Εάν δεν βρεθεί μια λύση σε αυτό, γνωρίζουμε ότι θα ξεκινήσουν συγκρούσεις για όλες, ανάμεταξύ όλων των μεγάλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε από πού θα χρειαστεί να γίνουν περικοπέ. Είτε πρόκειται για την κοινή αγροτική πολιτική, είτε πρόκειται για τα ταμεία συνοχή για, για τα πάντα θα γίνει χαμός. Ε, και το Και το δεύτερο λοιπόν μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει να δούμε είναι αν θα ενταχθεί το ΕΤΑ στον προπολογισμό, γενικό προπολογισμό. Ε, ούτε υποστηρίζω αυτό. Γιατί αυτό θα δώσει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παρατηρητή, ο οποίο όμω δεν έχει ουσιαστική δυνατότητα παρέμβαση. Εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη ενταχθεί στον προπολογισμό, τίθεται και το εξή ζήτημα. αυτή η ένταξη θα αυξήσει τους, τους συνολικούς πόρους που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή θα μειωθούν οι συνολικοί πόροι προς όφελος άλλων πολιτικών. Άρα και πάλι έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που δημιουργεί το Brexit. Συγκρούσεις για το ποιε πολιτικές επικρατούν ή είναι προτεραιότητες. Και πρέπει να δούμε λοιπόν πού λείπουν κατά κύριο λόγο, κατά μείζωνα λόγο, πόροι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία δεν επισημούν την αύξηση των πόρων, των ίδιων πόρων. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα επηρεαστούν όλες αυτές τις συζητήσει από τις εκλογές, όχι μόνο τις εθνικές, πιθανώς και τις περιφερειακές. Πάντοτε θα βρεθούν δικαιολογίε ή λόγοι για να μπλοκάρονται οι συζητήσει. Και εγώ ανησυχώ για όλα αυτά. Λοιπόν, για αυτού του λόγου πρέπει να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη και σαφή και ισχυρή θέση στο Κοινοβουλίο. Αλλά να έχουμε και συνέστηση των κινδύνων που, που, που, που, που μα περιμένουν σε αυτήν την ε, κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Πρώτα είναι η κυρία Χάουταλα και μετά είναι η κυρία Τόρνανο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούμπικ για το σχέδιο νομοδότησης. Φαντάζομαι ότι θα συμπληρωθεί. Δεν είναι ότι δεν συμφωνώ με κάτι, απλά θα ήθελα να υπάρξουν κάποιε προστίκε στο σχέδιο γνωμοδότηση. Αυτό που με ενοχλεί αυτέ τι μέρε είναι ότι πιστεύω πω η Κομισιόν ήδη σκέφτεται μια ριζική αναδιάρθρωση των οπτικών μέσων και εργαλείων. Και νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς. Προσπάθησα να ακούσω και σήμερα το πρωί και να ε, μιλήσω κι εγώ και να πω, να προειδοποιήσω κάπω ε, του συνάδελφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το επιχείρημα για μεγαλύτερη ευελιξία θα υπάρχει. Ναι, χρειάζεται ευελιξία, το ξέρω. Και είναι τόσο πολλέ οι ανθρωπιστικές κρίσει που ευελιξία χρειάζεται, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ. Μακροπρόθεσμοι στόχοι όμως, τι κάνουμε με αυτούς. Αν η Κομισιόν τελικά κάνει αυτό το μείγμα των μέσων και εργαλείων, κάνοντας πιο εύκολη τη χρήση και για μη σαφώς καθορισμένους σκοπούς, τι θα συμβεί στη νομική βάση. Αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει ήδη από τώρα. Φοβούμε δε ότι θα μπορούσε να γίνει και μια προσπάθεια την κατηγορία 3 εσωτερική ασφάλεια και κατηγορία 4 για τις ξέρεις δραστηριότητες να τις ε, να θολώσουν κάπως τα νερά και, να, και τις διασχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών. Εμείς ως Επιτροπή και το Κοινοβούλιο γενικά πρέπει να επιμείνουμε στις πολύ στοιχειώδεις βασικές απαιτήσει για το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και την επίτευξη των στόχων σε ό,τι αφορά τον ανθρωπιστικό προπολογισμό και το προπολογισμό για την ασφάλεια. Πολλά καλά στοιχεία περιλαμβάνει το σχέδιο του κ. Ρούμπιχ. Πράγματι, οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε χρειάζονται αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε αυτό. Βέβαια πρέπει να είναι συνεκτικές πολιτικές αναπτυξιακές, οι στόχοι και η σχετική ατζέντα γιατί όσοι θα πρέπει να έχουν εξορθολογιστεί και να καλύπτουν όλο το πλαίσιο και φάσμα των πολιτικών. Πρόσεξα σήμερα το, το Βρετανό συνάδελφο από το Westminster που ήδη μίλαγε για Βρετανία και Ευρώπη. Πόσο στενοχωρήθηκα γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι ένα θαύμα θα συμβεί. Στη... Στο μέτρο τη ανάπτυξης πρέπει Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνουν στο δυνατό πιο κοντά. Γιατί μοιραζόμαστε παρόμοιες ιδέες για την ανάπτυξη. Και σε ό,τι αφορά τις οροφές, ε, τα άνωτα τα όρια συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Θα αυξηθούν οι ανάγκες Και αν θέλει η Ευρώπη να παραμείνει εξωπρεπής, πρέπει να αυξήσει αυτά τα τα όρια. Ο Σαρλ Γκέρινς δεν ξέρω ακριβώς πώς το εξέφρασε, είπε ότι μπορεί να έχουμε κάποιες αναταραχές και πράγματι μπορεί να έχουμε τέτοια προβλήματα κλιματική αλλαγή. Ο Σπάνος Συνάλφος μίλησε για την ε, Βυρική Χερσόνησο και την επίπτωση που έχει κλιματική αλλαγή. Άρα μόλις στην αρχή βρισκόμαστε και πρέπει τον προπολογισμό να τον χρησιμοποιήσουμε πολύ σοφά για τους περιβαλλοντικούς στόχους και να αντισταθμίσουμε την έλλειψη αμερικανικών δεσμεύσεων αν θέλουμε να βοηθήσουμε να μετριαστούν οι αλλαγές του κλίματος. Πιστεύω όμως ότι η συζήτηση πρέπει να είναι πολύ ανοιχτή και ειλικρινή με την Κομισιόν για αυτέ τις νέες ριζοσπαστικέ ιδέες για το τι θα κάνουμε τα νέα εργαλεία. Η συζήτηση για τα μέσα θα έρθει λίγο αργότερα. Θα γίνει η πρώτη συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά θα δούμε τα μέσα ε, και πρέπει να συμμετέχουμε στην όλη συζήτηση έχει το λόγο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας και λαμβάνετε το λόγο. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είμαι καινούρια στην Επιτροπή σας και ελπίζω να μπορέσω να συνεργαστώ καλά με τους υπολείπους. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Ρούμπιχ για τη δουλειά του και ελπίζω ε, να μπορέσω να υποβάλω και τροπολογίες που θα εμπλουτίσουν το κείμενο. Όσον αφορά το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, σίγουρα είναι προφανής προτεραιότητα και θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για δέσμευση των κρατών πρωτίστως, αλλά και φορέων όπως οι επιχειρήσεις, ε, ενώσεις, ε, συλλογικά όργανα κλπ. Ε, οι δεσμεύσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ε, τις δεσμεύσεις των χωρών που είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει ε, να σεβαστούν αυτές τις δεσμεύσεις. Όσον αφορά την αύξηση της στήριξη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των στόχων αυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα κράτη πρέπει να αποφασίσουν πού θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε χρηματοδοτήσει, σίγουρα αιτιολογημένες, αλλά να δούμε και πόσο σημαντικές είναι. Θα πρέπει να επιμείνουμε στους στόχους που αφορούν το νερό, τη διατροφή, την υγεία αλλά και την παιδεία, ε, την εξυγίανση, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές. Όσον αφορά τις καινοτομίες και την ε, διακυβέρνηση ε, θα πρέπει να τα προωθήσουμε χωρίς όμως να χάσουμε και τους πιο επίγοντες στόχους. Ε, συμφωνώ με την ιδέα ότι η δημόσια ενίσχυση για την ανάπτυξη θα μπορούσε να διευκολύνει την κινητοποίηση ε, και άλλη χρηματοδότηση, γεγονό το οποίο θα επιτρέψει να αναπτύξουμε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων που πάντα επιθυμούμε. Όσον αφορά την ε, βοήθεια για ανθρωπιστική βοήθεια μετά από φυσικές καταστροφές, ε, ή ε, καταστροφές που προέρχονται από τον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να ε, κάνουμε να πληρώσουν αυτοί οι δράστες και όχι οι φορολογούμενοι των χωρών. Όσον αφορά την άξιση του προπολογισμού, νομίζω ότι δεν είναι αδόκιμο να λάβουμε υπόψη μας και το Brexit και το γεγονός ότι χάθηκαν κάποια στοιχεία δεν χρειάζεται να ε, εκμεταλλευόμαστε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι η ανάπτυξη για να ενοχοποιούμε το βρετανικό λαό ο οποίος έκανε ε, μια κυρίαρχη επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου κάποια πράγματα. Καταρχάς, το όλο θέμα ε, των στοιχείων εκτός προπολογισμού. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τη σύσταση αυτών των καταπιστευμάτων και νομίζω ότι ε, ε, θα μπορούσε να δικαιολογείται να έχουμε αυτά τα καταπιστεύματα εκτός προϋπολογισμού αν υπήρχαν κάποιοι εξωτερικοί φορείς που τα χρηματοδοτούν. Εάν όμως είναι εξωτερικά μέσα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε καταπιστεύματα για τα οποία δεν υπάρχει δημοκρατική εποπτεία. Ε, πέραν αυτού, στο σημείο 5 στην έκθεσή σας ε, για το ε, συμπερίληψη του ΕΤΑ στον προπολογισμό, ε, νομίζω ότι η ανησυχία μου είναι αυτή που έχετε στο τέλος. Ε, η συμπερίληψή του στα πλαίσια της συνολικής αύξησης ε, των ε, συνόλου των ε, στόχων της που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχουμε κάποια εγγύηση, δεν είναι λογικό να ενταχθεί στον προπολογισμό, γιατί τότε μπορεί να φαίνεται ότι αυξήθηκε ο προπολογισμό, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να έχουμε σημαντικές περικοπές, που με φτάνει και στη συζήτηση για τον Brexit. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το θέμα δεν είναι να κατηγορούμε αλλήλους, απλώς να αναφέρουμε γεγονότα. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλει περίπου το 50% ε, του ΕΤΑ, που σημαίνει ότι είναι περίπου 5 δις ευρώ και το 10% του TCIA και αυτό είναι συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου. 700 εκατομμύρια λίρες ε, από την ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν φύγει λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια πόλη στον προπολογισμό, αυτή ανέφερε και ο Σαλ Γκέρενς και είναι απλώς περικοπή στη χρηματοδότηση. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ελπίζω ότι μετά τα Χριστούγεννα θα έχουμε συμφωνία για να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Θα υπάρξει δηλαδή μια συμφωνία και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Και μπορεί και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι μεγάλος χορηγός τη ανθρωπιστική βοήθεια, ε, έχει 1,7%, το 0,7% ήδη στην ομοθεσία του, ίσως να συνεχίσει να συνεισφέρει. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, δεν ξέρω τίποτα για την κυβέρνηση, απλώς η άποψη προσωπική μου είναι ότι είναι λογικό να συνεχιστεί. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα του ΕΤΑ, αλλά θα μπορούσε ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει και μια χειρονομία καλή θελήσεω ε, το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση. Πρέπει να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και να ακούσουμε και την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το κρίσιμο ζήτημα θα είναι τα ανώτατα όρια. Γιατί αυτό ξεκινάει το 2021. Είναι ο προπολογισμό για του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μόλι τελειώσουν αυτέ οι δημοσιονομικέ ε, ε, ε θα έχουν τελειώσει η περίοδος των στόχων της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Θα είμαστε ήδη στο 2028 και θα πρέπει να τους έχουμε επιτύχει. Δεν βλέπω κάποιον να ζητά το λόγο. Έχουμε και εκπρόσωπο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ακούσουμε και την άποψή της λοιπόν. Um, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας όσον αφορά αυτό το προσχέδιο νομοδότησης και αυτά που ακούστηκαν στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι αυτό το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για να σκεφτούμε και να αντικατοπτριστεί τι αυτό στο πολιετές πλαίσιο ε, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη και το θεματολόγιο 2030, αλλά εγώ επίση θα αναφέρω και τη συμφωνία τη ε, Αντισα... Άμπαμπα και ε, στην οποία επαναβεβαιώσαμε την δέσμευσή μας για το 0,7% του ΑΕΠ και επίσης, και εξίσου σημαντικό, το 0,2% για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Επομένως, για να πετύχει κανείς αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί συλλογικά, δεν ε, μπορεί να συμβεί αυτό μόνο με την ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το, το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με την συνεισφορά των κρατών μελών. Το επόμενο λοιπόν πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κατά την άποψή μου ένα, ένα εργαλείο για να καταλήξουμε ότι συνεχίζουμε να, έχουμε, να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτούς τους στόχους. οι οποίοι έχουν ε, μεταφραστεί και στην κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ε, η συζήτηση για την ένταξη στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη. Η έκθεση τονίζει το ύψος του πιστώσεων, το ύψος του ταμείου και πού θα τεθεί το ανωτοτόριο. Ε, δεν είναι δεδομένο ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα συμφωνούσαν στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας. Η συζήτηση αυτή ε, θέτει και κάποια άλλα ζητήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα του αποθεματικού ή γενικά των αποθεματικών, που αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας με το ΕΤΑ. Και γενικότερα το, το ζήτημα της ευελιξίας με, στη χρήση του ΕΤΑ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό του ποθεματικού ήταν της τάξης του 20%. Αλλά και αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό ε, θετικό στοιχείο του τρέχοντος ΕΤΑ. Ε, γιατί ε, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιποκρινόμαστε στις αλλαγές και στις μεταβολές που πολιτικών προτεραιοτήτων που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πολιετού πλαισίου. Έχουμε ήδη δει ότι δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα στην αρχή του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό το αποθεματικό μας έδινε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε. Εάν λοιπόν το ΕΤΑ ενταχθεί στον ε, προϋπολογισμό, τον ιδρικό, το ζήτημα που θα τεθεί είναι τι θα γίνει και με το αποθεματικό του. Πώς θα ενταχθεί το αποθεματικό στον, στον γενικό προπολογισμό. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να στο οποίο θα θέλει να προβληματιστούμε είναι το ότι οι τρέχουσες μορφές εξόδων που καλύπτονται από το, ε, σημαντικό, ε, το σημερινό ΕΤΑ ίσως να μην μπορούν να συμπεριληφθούν για νομικούς λόγους στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Το οποίο αμέσως θα δημιουργήσει πρόβλημα θα τεθεί το ζήτημα του τι θα γίνει με αυτές τις πιστώσεις, με αυτά τα έξοδα και τι θα τις αντικαταστήσει, τι είδους εργαλείο θα μπορούσε να αντικαταστήσει για παράδειγμα τις πιστώσεις για δράσεις ε, ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχει επίση και η γενικότερη συζήτηση που αναφέρατε για την αρχιτεκτονική, για τη δομή των διαφορών χρηματοδοτικών μέσων. Ενώ υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής, διεθνές και μετά ευρωπαϊκό, σήμερα έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά εργαλεία για την χρηματοδότηση. Στο σύνολό τους είναι 15, με 15 διαφορετικές νομικές βάσεις και ε, σκεφτείτε το εξής αυτή τη στιγμή για το, στο, κεφάλαιο, στον τίτλο 2 έχουμε έξι φορές το ποσό του τίτλου 4 και μικρότερον αριθμό εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων. Επομένω έχει υπάρξει αυτή ο άναρχος πολλαπλασιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων ε, που ισχυρίζομαι και ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της ε, αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμπτύξουμε τα εργαλεία όπου χρειάζεται, ε, λαμβάνοντας υπόψη μας την φύση που θα έχουν τα, τα προγράμματα αναπτυξιακής ε, βοήθειας που θα αναλάβουμε στο πλαίσιο του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, αυτό δεν περιορίζει ή δεν υπαγορεύει κάποιες διαφορετικές επιλογές όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική της πολιτική. Αυτούς τους προβληματισμούς που θέλω να μοιραστώ μαζί σήμερα. Ξαναδώσω τώρα το λόγο, λοιπόν, των Παύλο Ρούμπιχ. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω θερμό όλου τους συναδέλφους για τι παρατηρήσει πάρα πολύ χρήσιμε για μένα. Νομίζω ότι πολύ απλά αυτό που είπατε είναι ότι και στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να βρούμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, που δηλαδή μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει προσθέμενη αξία σε σχέση με την εθνική, ε, εθνικώ προσφερόμενη αναπτυξιακή βοήθεια και σίγουρα και στο εθνικό επίπεδο ε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία δεν ε, υπάρχει πρόοδος και μπορούμε και πάντα στο πλαίσιο της επικουρικότητας κάτι να κάνουμε και σε ό,τι αφορά το Brexit εγώ μπορώ να δω και μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια νέα συνεργασία σε νέες βάσεις ε, και με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένες βάσεις θα πρέπει να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα οικονομικά. Και η επιθυμία θα ήταν οι πληρωμές των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να ληφθούν υπόψη, να συμπεριληφθούν. Η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί να ξεφύγει τόσο εύκολα με μια πληρωμή, γιατί οι πληρωμές που πρέπει να κάνει ε, πηγαίνουν ε, σε ένα μακρινό χρονικό ορίζοντα, καλύπτουν ε, πολλές ε, χρονιές. Και θέλουμε να δώσουμε μια νέα ευκαιρία στην αναπτυξιακή πολιτική. Δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, θα εργαστούμε από κοινού, θα υποστηρίξουμε μαζί ενωμένοι αυτές τις γραμμές, αυτές τις θέσεις. Έχουμε ένα κοινό στόχο και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου να έχουμε έναν καλύτερο ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω. Τι ψάχνω. Τις προθεσμίες τροπολογιών ψάχνω. Κέιτι, μήπως θέλεις κάτι να πεις στο μεταξύ. Ναι, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση της Κομισιόν. Δεν λέω ότι είναι λάθος να γίνει streamlining, εξορθολογισμό των μέσων. Αλλά θα πρέπει να γίνουμε πολύ προσεκτικό τρόπο. Αν δηλαδή στόχος είναι πραγματικά να είναι αποτελεσματική αναπτυξή πολιτική, δεν μπορεί να γίνει αυτό με κάποιο τυχαίο τρόπο. Δεν ξέρω αν πολύ σύντομα η Κομισιόν θα μπορούσε ακόμη να μας πει αν υπάρχει κάποια ανάλυση, μελέτη αντικτύπου που έχει ξεκινήσει. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Ναι, έλεγα ότι θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν εάν έχει ξεκινήσει μια μελέτη αντικτύπου και αν θα συμμετέχει η Επιτροπή μας και γενικά το Κοινοβούλιο σε κάποιες πρόορες συζητήσεις ίσως. Κομισιόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο πρόγραμμα εργασίας του χρόνου για την Κομισιόν έχουμε μια πρόταση το Μάιο του χρόνου για το πολιτές πλαίσιο και κατά πάσα πιθανότητα ταυτόχρονα ή λίγο μετά θα κατατεθούν προτάσεις για τα νέα μέσα. Σε πλήρη σεβασμό με την ε, προσέγγιση για καλύτερη νομοθεσία. Έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο τη ενδιάμεσης αναθεώρησης ε, των μέσων οι εξολογήσεις, έχει γίνει και δημόσια διαβούλευση και θα γίνει και μελέτη αντικτύπου που θα δημοσιοποιηθεί από κοινού με την πρόταση της Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι στην όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν ευκαιρίες σε διαπλήσεις με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 6 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, 6 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 24 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστούμε τον Παλουρούμπιχ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περνάμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, το σημείο 14, ανθρωπιστική κατάσταση στην Καραϊβική μετά τους πρόσφατους τυφώνες. Έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές, ε, τους οποίους ε, θα φέρουμε εδώ στο πάνελ. Ένα λεπτάκι διάλειμμα λοιπόν για να έρθουμε εδώ στο Προεδρείο. Okay, colleagues, we're moving on to item 14. Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 14, όπως είπα είναι πολύ σημαντικό σημείο. Παρακαλώ όσοι αποχωρούν, παρακαλώ λίγο ησυχία. Υπάρχουν πολλοί που βλέπουν στο διαδίκτυο, το ξέρω, γιατί έλαβα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κόσμο που ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Είχαμε τυφώνες στην περιοχή της Καραϊβικής, είχαμε τον τυφώνα Ήρμα και μετά τον τυφώνα Μαρία. Και κάποιες ε, χώρες λοιπόν ε, καταστράφηκαν όλος ε, ξέρω ότι στο Σαμαρτάν, στις Γαλλικές Αντίλες το 95% της επικράτειας καταστράφηκε. Και ορισμένες φορές αναφερόμαστε σε αυτές τις καταστροφικές φυσικές θεομηνίες. Τη μια εβδομάδα είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα και μετά εξαφανίζεται. Αλλά εμείς θέλουμε να παραμείνει στην επικαιρότητα γιατί γνωρίζουμε από διμερείς επαφές ε, τι συνέβη στην Καραϊβική και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που της αναλογεί για να αποκαταστήσει αυτές τις περιοχές. Ε, αυτά τα νησιωτικά κράτη. Σήμερα γίνεται μια πολύ μεγάλη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη και ξέρω ότι είναι και ο Επίτροπος εκεί ε, είναι λοιπόν πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή αλλά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας, ένας, ε, μια περιοχή με την οποία έχουμε ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς ε, και φυσικά κάποια είναι και τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χαιρόμαστε λοιπόν εδώ που έχουμε εκπροσώπους ε, των χωρών της Ανατολικής Καραϊβικής και έχουμε και εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Θα ξεκινήσω όμως με την κυρία Σαρλίν Σίγκλφορντ Μακκλίμον που είναι η ομιλήτρια εκ μέρους της Καραϊβικής που είναι η επικεφαλής ε, των πρεσβειών ε, των χωρών της Ανατολικής Καραϊβικής και των αποστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι εκπροσωπείτε μια σειρά από χώρε. Μπορείτε να μα εξηγήσετε εσεί ποιου εκπροσωπείτε και καλό θα ήταν να μα παρουσιάσετε εσεί μια εικόνα του που βρισκόμαστε σήμερα, ε, το επίπεδο του προβλήματο και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για την ε, κατεπίγουσα βοήθεια και τη Γενική Διεύθυνση ε, ΔΕΦΚΟ για την διάσκεψη που γίνεται σήμερα και τι μπορούμε να περιμένουμε για μακροπρόθεσμη υποστήριξη. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και για την πρόσκληση να μιλήσω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα και πραγματικά θα ήθελα να σας φέρω και θερμούς χαιρετισμού από την Καραϊβική παρά και το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο καιρός μας δεν ήταν και τόσο ε, ε, πρόσδεκτος. Εκπροσωπώ τέσσερις χώρες της Ανατολικής Καραϊβικής ε, στο Βέλγιο αλλά στην Καραϊβική είμαστε τμήμα της οργάνωσης των χωρών της Ανατολικής Καραϊβικής που περιλαμβάνει 10 χώρες και μη ανεξάρτητες χώρες, τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Μαρτινίκα που είναι υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας. Το θέμα των τυφώνων στην Καραϊβική είναι κάτι το οποίο βλέπουμε υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, επομένως θα σας μιλήσω και για τον αντίκτυπο και από αυτή την ε, οπτική γωνία, την κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο που είχε για το χρέο μας και για τη ε, συνεχή ευάλωτη κατάστασή μας. Όπως γνωρίζετε, διότι ήταν και στην επικαιρότητα και ξέρω ότι θα μιλήσει η Γενική Διαθεσία ΕΚΟ για την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, δεν ε, θα σα μιλήσω για αυτά, θα σα πω τι βιώσαμε εμεί. Είμαστε μια ζώνη υψηλού κινδύνου, είμαστε κάθε χρόνο σε κίνδυνο, Συνεχώ από τροπικέ καταιγίδε, τυφώνε, πλημμύρε, ξηρασία, ανύψωση του επίπεδου της θάλασσας και απώλεια της ακτογραμμές. Είμαστε νησιωτικά κράτη και κάποια από τα νησιά μας χάνουν ε, τμήμα της ακτής κάθε χρόνο. Χάνονται στον ωκεανό, καλύπτονται από τον ωκεανό και επομένως είμαστε συνεχώς ευάλωτοι. Εγώ είμαι από τη Δομήνικα, ε, η οποία επλήγει... Ε, από τον τυφώνα Μαρία όταν μόλις είχαμε αρχίσει να ανακάμπτουμε από την ε, τροπική καταιγίδα Έρικα. Ε, η οποία κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερό το νησί. Και αυτό ήταν απλώ ε, μια απλή βροχόπτωση. Και ο λόγο που μα επηρέασε τόσο πολύ μια βροχόπτωση ήταν γιατί είχαμε μια συνήθιστη περίοδο ξηρασίας. Συνήθω δεν έχουμε. Είμαστε ένα τροπικό ορεινό νησί και υπήρχε μια μεγάλη ε, περίοδο ξηρασίας. Ήρθε η βροχή η οποία έπεσε απευθεία στη θάλασσα μετά από τόσο μεγάλη ξηρασία. Μόλι είχαμε αρχίσει να ανακάπτουμε, τα πηγαίναμε καλά και όταν χτυπήθηκαν η Αντίγουα και τα Μπαρμπάντο ήταν πολύ ισχυρό το χτύπημα εκεί, κυρίω στην Αντίγκουα. Κάποια από τα διδάγματα που αντλήσαμε και κάποια προετοιμασία ήταν να αποθηκεύσουμε περαιτέρω τρόφιμα, τα οποία στείλαμε στην Παρμπούντα και σε άλλα νησιά τα οποία επλήγησαν και είχαν χάσει ε, όλες τους τις προμήθειες. Όπως θα γνωρίζετε, η Παρμπούντα αυτή τη στιγμή είναι κατοίκητη και είναι η πρώτη φορά σε 300 χρόνια που δεν υπάρχει κάτοικος ε, στο νησί. Και βεβαίω, ε, μετά από μια εβδομάδα που στείλαμε τι προμήθειε μα, μα έπληξε ο τυφώνα Μαρία και βρεθήκαμε ανυπεράσπιστοι ε, γιατί δεν μπορούσαμε να ε, θρέψουμε τον πληθυσμό μα μετά από το χτύπημα του τυφώνα αλλά είμαστε και πλήρω ανυπεράσπιστοι και σε όλα στι άλλε πτυχέ. Όσον αφορά λοιπόν την κατάσταση τη Καραϊβική αυτή τη στιγμή το μόνο ερώτημα είναι ποιο νησί δεν επλήγει. Έχουμε πάνω από 17 νησιά τα οποία επλήγησαν και από τον τυφώνα Μαρία και από την Ήρμα και αυτό αφορά όλες τις ε, ε, υπερπόντιες περιοχές ε, των κατοχωρών, τη Γαλλία, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και φυσικά και την ανεξάρτητη Καραϊβική. υπάρχει και κάτι το οποίο θεωρώ προτεραιότητα στη συζήτηση αυτή συνολικά. Μεταξύ του 1990 και του 2017 η Καραϊβική επλήγει από 320 φυσικές καταστροφές και αυτό είχε ε, κατά συνέπεια 13 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους ε, στην περιοχή της Καραϊβικής. Είναι μία από τις πιο υπερχρεωμένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή έχουμε με χρέος 49 δισεκατομμύρια, αλλά τα 31 δισεκατομμύρια αφορούν φυσικές καταστροφές, ανοικοδόμηση κλπ. Και να σας το εξηγήσω λίγο αυτό. Γνωρίζετε ότι εμείς θεωρούμαστε χώρες μεσαίου εισοδήματο βάσει του κατακεφαλήνα ΕΠ που είναι κάτι για το οποίο διαμαρτυρέμαστε συχνά γιατί δεν είναι λογικά αν μπορεί να καταστραφεί ένα ένα νησί ολόκληρο σε τέσσερις ώρες, πώς μπορεί να σε χώρα μεσαίου με εισοδήματο και να χάνει όλη την ανθρωπιστική βοήθεια. Και παρακολούθησα και τι άλλε συζητήσει και από τα άλλα θέματα μπορεί να είναι χρήσιμο να γνωρίζετε αυτέ τι πληροφορίε και να συνεχίσετε το διάλογο ε, και χωρί τη δική μα τη φωνή. Ε, λοιπόν, τα 31 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια αφορούν την ανοικοδόμηση, γιατί κάθε φορά δεν καταστρέφεται πλήρως ένα νησί, παίρνουμε ένα δάνειο για να ξανακατασκευαστεί ένα ε, λιμάνι, ε, για παράδειγμα, στο Κίτσε Νέβης που χτυπήθηκε από τον τυφώνα Μαρία, υπήρχε μια μαρίνα η οποία πρόκειται να ανοίξει και καταστρέφηκε ολοσχερός. Δεν μπόρεσε να γίνουν καν τα εγγένεια, αλλά φυσικά πρέπει να την αποπληρώσουμε και να την ξαναχτίσουμε. Και ε, αυτό είναι αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Χάνουμε υψηλό εισοδήμα, τα χάνουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση, την προνομιακή χρηματοδότηση, αρχίζει η ανοικοδόμηση και μετά χτυπάει ένα τυφώνα στην επόμενη χρονιά και τα ξαναρχίζουμε όλα από την αρχή. Πρέπει να το έχετε και κατά νου. Ε, είμαστε πολύ ευάλωτοι και μάλιστα ε, αυτή η διαδικασία είναι συνεχής. Δεν σταματά ποτέ αυτή η ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Σας είπα λοιπόν για ποιο λόγο υπάρχει το χρέος στην περιοχή μας και ε, θα ήθελα εδώ να μοιραστώ μαζί σου και αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχουν 10 χώρες που υπερβαίνουν το 60% χρέους του ΑΕΠ δύο που υπερβαίνουν το 220 και τέσσερις που υπερβαίνουν το 90%. Αυτή είναι η κατάσταση στην Καραϊβική και πρέπει να ξαναχτίζουμε συνεχώς. Και σας τα λέω αυτά διότι αποδεικνύουν πόσο πολύ ε, εξαρτόμαστε και πρέπει να εξαρτώμαστε από τους εταίρους μας για την ανοικοδόμηση και για την ε, κατεπίγουσα βοήθεια. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να τα ξέρετε. Επίσης συμμετέχουμε σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για το θέμα του τι θα γίνει μετά το κοτονού. Υπάρχουν πολλές ε, χώρες, πολλές από αυτές είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και δεν έχουν καν το χρέο που διαθέτουμε εμεί σε αυτές οι χώρε. Ξέρουμε ότι 38 χώρε στην υποσιοχάρη Αφρική έχουν μόνο 59% ε, χρέος. Ε, η Ινδονησία επίση είναι στο 55%. Εμεί υπερβαίνουμε το 100% και έχουμε 10 χώρε που υπερβαίνουν το 90%. Άρα βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, για να επανέλθω αυστηρά στο θέμα των τυφώνων τι έγινε φέτος το φθινόπωρο στο Σεπτέμβριο. Είχαμε δύο τυφώνες κατηγορίας 5 μέσα σε δύο εβδομάδες. Αυτή είναι κατάσταση η οποία δεν έχει ε, ξαναπαρουσιαστεί. Είχαμε τον τυφώνα Μαρία που αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Σε λιγότερο από 13 ώρες πέρασε από ε, κατηγορία 1 σε κατηγορία 5 και ε, συνήθως ε, τα σπίτια μας αντέχουν στην κατηγορία 3, μπορεί και κατηγορία 4, αλλά εδώ είδαμε εκτεταμένες ζημιές σε σχεδόν όλα τα σπίτια. Πάνω από το 90% των υποδομών καταστράφηκε στη Δομήνικα, ε, τα πάντα εξαφανίστηκαν στην Παρμπούντα, στο Σαν Μαρτάν ε, δεν, έχουν, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά δεν ε, αλλάζει ε, η εθνικότητα τους ανέμους. Όταν χτυπάει ο άνεφος ε, παρασύρονται τα πάντα. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το σπίτι των γονιών μου δεν έχει στέγη και κάποια σπίτια απλώς μετακινήθηκαν. Ολόκληρα κομμάτια γης αποσπάστηκαν, σπίτια κατέληξαν στην όχθη. Ε, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. 95% είναι χωρίς ρεύματα, συστήματα υδροδότησης ακόμα είναι προβληματικά και οι περισσότεροι είναι άστεγοι. Ε, και το ίδιο θα συμβαίνει και στις παθένες νήσους ε, τις Βρετανικές, ε, το Σαμαρτάν επίσης, σας είπα η Μπαρμπούντα για πρώτη φορά σε 300 χρόνια είναι ακατοίκητη. Και οι συνέπειες για μας, αν θα μπορούσα να σας πω και κάποια πράγματα, είναι ότι το 90% των υποδομών μας καταστράφηκε, 100% της γεωργίας μας στέγαση, παιδεία, ε, αλληλεία, δασοκομεία. Το θέμα των δασών είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλά νησιά της Καραϊβικής ε, έχουν αγροτουρισμό, πεζοπορίες, καταδύσεις. Ε, το νησί καταγωγής μου, η Δομήνικα, θεωρείται το νησί της φύσης της Καραϊβικής και εμείς προστατεύουμε τα δάση μας μέσω νομοθεσίας και ε, ο θαλάσσιο περιβάλλον. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά είναι από τα εθνικά μας ε, πάρκα εδώ και 20 χρόνια είναι πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Δεν έχουμε διεθνές αεροδρόμιο, δεν έχουμε αλυσίδες ξενοδοχείων, δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Έχουμε δύο μεγάλα ξενοδοχεία για τα στάνταρ της Καραϊβικής, αλλά τα περισσότερα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρή ξενώνας. Δεν κόβουμε δάση για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και ε, μάλιστα ε, θεωρούμαστε ε, και ότι συνεισφέρουμε στην μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη ακριβώς όσοι επειδή προστατεύουμε τα δάση μας και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή ε, στον πόλεμο για την κλιματική αλλαγή και ο Πρωθυπουργό μας το είπε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο και το είπε και στη Βόνη την προηγούμενη εβδομάδα. Οι χώρες της Καραϊβικής δεν έχουν ε, συμβάλει καθόλου στην κλιματική αλλαγή, στις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Δεν μπορούμε καν να πούμε ότι άλλαξε καθόλου δείκτης χάρη στη συμβολή μας. Ε, και ε, αυτή τη στιγμή είμαστε κατεστραμμένοι και είμαστε και ανίκανοι να κάνουμε το οτιδήποτε. Γι' αυτό ακριβώ και αναζητούμε εταιρική σχέση με χώρε τη Ευρώπη και άλλε χώρε. Ο αντίκτυπο για μα είναι κοινωνικό, είναι ανθρώπινο, είναι οικονομικό, έχουν κλείσει επιχειρήσει, ε, ε, διακόπηκε η οικονομική δραστηριότητα, χάθηκαν θέσεις εργασίας, ε, τουρισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί, έχουμε και ε, ασθένειες λόγω μολυσμένου νερού, κατεπίγουσα κατάσταση στις ιατρικές υπηρεσίες. Είναι γνωστό ότι έχουμε την υψηλότερη συγκέντρωση ατόμων άνω των 100 ετών ε, και πεθαίνουν όχι από τον τυφώνα, αλλά από τις συνέπειες του τυφώνα, γιατί δεν υπάρχει ιατρική υπερίθαλψη. Ε, δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε ε, φάρμακα, δεν μπορέσαμε να τα αποθηκεύσουμε. και υπάρχουν ανθρώπινες λοιπόν και οικονομικές συνέπειες, αλλά και το θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό. Η Καραϊβική είναι περιοχή διέλευσης ναρκωτικών, όπως γνωρίζετε, από το βορρά προς τον νότο, ε, συγγνώμη, από νότο προς το βορρά. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ελέγχουμε την κατάσταση κατάσταση, επομένως ε, ε, και η ασφάλεια των συνόρων μας ε, πλήττεται. Και φυσικά πολύ λυπηρό για μας έχει καταστραφεί η βιοποικιλότητα, διότι ένα στα εκατό δέντρα έμεινε όρθιο και φυσικά και η χλωρίδα και η πανίδα έχουν πληγεί και βρισκόμαστε ήδη στον κατάλογο των χωρών που έχουν μεγάλο κίνδυνο εξαφάνισης ειδών από τη βιοπικιλότητα και αυτή είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ, ε, διότι όπως είπα ξέρω ότι η Γενική Διευθυνσία ΕΚΟ θα μιλήσει για την ανθρωπιστική βοήθεια που λάβαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά θα ήθελα να σας πω κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να γνωρίζετε για το πόσο ευάλωτοι είμαστε, το γεγονός ότι έχουμε υποπέσει ένα φαύλο κύκλο που χτίζουμε και ξαναχτίζουμε συνεχώς, θεωρούμαστε χώρες ε, μεσαίου ε, εισοδήματος, αλλά θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στις παρυφές αυτών των εξισώσεων. Δεν μπορούμε να θεωρούμε Ε, ε, Χώρε υψηλού εισοδήματο πρόκειται να μπει αντίγκο στον κατάλογο και καταστράφηκε σε μερικέ ε, ώρε ε, το νησί. Τι υψηλό εισόδημα είναι, τι μπορούμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη όταν είναι τόσο ευάλωτα τα πράγματα και είναι τόσο περαστικά. Ε, μας ανησυχεί το υψηλό χρέος, το οποίο όμως έγινε σε 35-40 χρόνια και αφορά και πάλι την ανοικοδόμηση. Το γεγονός ότι πρέπει να ανοικοδομήσουμε με ίδιου πόρου ή με δάνεια, γιατί θεωρούμαστε οι μεσαίου εισόδηματο. Ε, δήματος και έχουμε και το φορολογικό περιθώριο να το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες και ε, συνεχίζει όσα τα θέματα και εμείς θεωρούμε ότι είναι ε, μη ρεαλιστικό και ευχαριστούμε τις χώρες της Ευρώπης που μίλησαν στον ΩΣΑ και ε, δεν νομίζω ότι ήταν μάταιη η συζήτηση. Κάπου θα οδηγήσει όλη αυτή η συζήτηση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας πω κάτι που είπε ο Πρωθυπουργό στη Βόνη την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και δεν είναι μεταφορικό αυτό ο ε, ε, πόλεμος, ούτε μεταφορική γραμμή. Είναι μια γραμμή στην οποία θάβουμε τους νεκρούς μας. Ε, τρέφουμε τις φλιγές μας και ζητάμε ενισχύσεις. Και με αυτό Νομίζω ότι θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ, εκτός και αν έχετε ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την περιγραφή της κατάστασης. Για τους συναδέλφους που δεν ήταν παρόντες, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ότι για πρώτη φορά μετά από 300 χρόνια δεν υπάρχει ε, ψυχή στο νησί Μπαρμπούντα. Ναι, Έχω επισκεφθεί την Ντομίνικα πρόσφατα σχετικά και είναι ε, εξαιρετικά λυπηρό. Τραγικό πω μεγάλε καταστροφέ υποστήκατε και πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι τοπικέ κοινότητε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη ε, ΕΚΟ, τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστική Βοήθεια, ο κύριο Λάντκραφ. Ε, αν μπορείτε κάπω να μην μακροβολήσετε, να μα δώσετε τα κύρια σημεία για να έχουμε τη δυνατότητα να γίνει και η συζήτηση στην Επιτροπή. Κύριο Λάντκραφ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η... Λάντκραφ και είμαι διευθυντής ειδικά για το τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας που ασχολείται με την Καραϊβική. Θα προσπαθήσω να ε, σας περιγράψω την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την ε, κρίση, η οποία ήδη περιγράφηκε πολύ αναλυτικά. 5 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν, και οι υλικέ ζημιέ ε, όσον αφορά τι κατοικίε, ε, το, τον ηλεκτρισμό, το νερό, την αποχέτευση ήταν επίση πολύ σημαντικές. Ποια ήταν η ανταπόκριση. Ίσως να γνωρίζετε ότι το κέντρο συντονισμού για έκτακτες ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας παρακολουθεί τις καταστάσεις αυτές σε όλο τον πλανήτη σε 24ωρη βάση και παρακολουθήσαμε από κοντά τις ε, ε, κινήσεις ε, των τυφώνων. Επομένω προετοιμαστήκαμε με ειδικού, με πυρογνώμονε που ήταν έτοιμοι να επισκεφτούν το νησί για να αξιολογήσουν την κατάσταση και δεν ήταν εύκολο να έχει κανείς πρόσβαση σε όλα τα νησιά ιδιαίτερα εξαιτία κατά τη διάρκεια του τυφώνα Μαρία. Έγιναν βέβαια και διάφορε συναντήσει συντονισμού με κρατη δεν θα μπω στι λεπτομέρειε τώρα σε αυτέ, γιατί το ζήτημα είναι να δούμε τι τελικά παρήχαμε στι χώρε αυτέ. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, εξοπλήθηκαν περίπου, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι διαθέσιμα, ε, σταδιακά, καμιεύτηκαν. Αξιοποιήσαμε το Ταμείο τη Διεθνή Επιτροπή Ρηθρού Σταυρού για την ανταπόκριση στι ανθρωπιστικέ καταστροφέ. Υπήρξε επίση χρηματοδότηση από την Κούβα, από τον Άγιο Μαπίνο, από την Δομήνικα. Και η Αντίκου και η Βαρμπούντα ήταν ε, και η οι κυρία αποδέκτε. Δημιουργήθηκαν καταβλισμοί προσωρινή 65.000 ατόμων από τον ΟΗΕ και 25.000 μετά από συντονισμό με την κυβέρνηση και μετά από αυτόν τον συντονισμό με την κυβέρνηση υπήρξαν περιοχές που ποσών κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Αξιοποιήθηκε επίσης ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση της Ντομίνικα μια ομάδα ειδικών πολιτικής προστασίας πήγε στο νησί για να βοηθήσει την, ε, τον συντονισμό με εκπροσώπους πολλών κρατών μελών από τη, την Ολλανδία, τη Γαλλία, της, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, συνεισέφεραν επίσης με συστήματα καθαρισμού του πόσιμου νερού, ε, με σκηνές, με ταμπλέτες για τον καθαρισμό του νερού και τέτοιου τύπου ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ η ανταπόκριση. Αυτή είναι η γενικέ γραμμέ η ανταπόκριση που είχαμε. Θα μπορούσα να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε και να των ερωτήσεων, το επιθυμείτε. Το σημαντικό πάντω από τη δικιά μα την πλευρά είναι ότι είχαμε πολύ καλό συντονισμό ε, με του συναδέλφου που ασχολούνται με τα ζήτηματα τη αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, έτσι ώστε όταν τελειώσει η άμεση ανταπόκριση στην κρίση να υπάρξει μια ομαλή μεταβατική ε, περίοδος, μια μετάβαση στην πιο μακροπρόθεσμη δουλειά που θα χρειαστεί. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ε, ευτυχές που μπορέσαμε να το καταφέρουμε. Και τώρα σιγά σιγά περνούμε πλέον σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στην Κούβα ήταν εκείνη που χρειαστήκαμε περισσότερο να επέμβουμε άμεσα με τροφή και νερό, δευτερευόντως όπως είπα στην Αντίγουα Βεβούντα. Και με την αδειά σα, κύριε Πρόεδρε, να δώσω το λόγο στου συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξική Συνεργασία για να σα πούν πώ αντιμετωπίζουν το ζήτημα από τη δικιά του την πλευρά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι είναι σημαντικό να ακούσουμε και από την ΓΔ Ντεύκο. Ευχαριστώ. Καρλίνα Αντρέας λέω. Και είμαι η αναπληρωτρία τομεάρχης με τη συνεργασία με Λατινική Αμερική Καραϊβική. Είναι σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Επιτρόπο Μίμητσα. Παρίσταται στην ε, διάσκεψη ψηλού επίπεδου των ε, χρηματοδοτών από την Κάρικομ και τα Ηνωμένα έχει οργανωθεί αυτή η διάσκεψη για να βελτιωθεί η αντοχή των πληγήσεων χωρών της Καραϊβικής από τους τυφώνες. Ε, στις 3 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης ήταν αυτή η συνεδρίαση για την χρηματοδότηση, 6 ώρες διαφορά. Ο Επιτρόπος θα ανακοινώσει ένα πολύ σημαντικό πακέτο χρηματοδότησης, 300 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ε, από την πλευρά της Ένωσης ε, για την βοήθεια που θα πρέπει να παρασχεθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών και την κάλυψη των προτεραιοτήτων στις πληγήσεις περιοχές μετά τους ε, τυφώνες. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση οικονομική που περιλαμβάνει τον επαναπροσανατολισμό και την προσταβαρή διάθεση για την ε, εφαρμογή προγραμμάτων. Έχουμε επίσης επιταχύνει κάποιες πληρωμές όπως και την υλοποίηση και την έγκριση νέων προγραμμάτων. Θα περιλαμβάνει το πακέτο αυτό όμως και σημαντική υποστήριξη ύψους 60 ε, εκατομμυρίων θα είναι νοπό χρήμα από τα αποθεματικά του 11ου ΕΤΑ. Συνολικά, το πακέτο μέσο και μακροπρόθεσμα, πακέτο υποστήριξη οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνάδελφοι από το ΕΚΟ να εφαρμόζουν. Άρα η μέσο μακροπρόθεσμη βοήθεια θα εστιάσει σε δύο τομεί. Δίμερε επίπεδο καταρχά, για να υποστηριχθούν ε, οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο, δηλαδή Δομήνικα, Σεν, Κιτσενέβη, Σαντίβα Μπαρμπούδα ε, και Κούβα, για μακροπρόθεσμη ανάκαψη και ανοικοδόμηση, βασικές υπηρεσίες και επανάληψη των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτή και κάποια άλλη βασική στόχη. Δεύτερη προσέγγιση, σε περιφερειακό επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση θα Θέλει ε, με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια αντοχή μακροπρόθεσμη, ανθεκτικότητα μακροπρόθεσμη και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το δούμε από το περιφερειακό πρίσμα. Ενίσχυση διαφόρων θεσμών ε, και οργανισμών που απέδειξαν άκρος αποτελεσματική και αμέσως μετά την καταστροφή σε η Management Agency. Αυτό σημαίνει το ακρονίμιο. 14 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση αυτού του φορέα προβλέπουμε για το πώς μπορεί να είναι πιο αφεκτική περιοχή. Αυτό θα μας απασχολήσει και πώς θα εξελισσόμαστε συνεχώς. Όπως και η κυρία Μακίλμουν. Για να μην ξαναρχίζουμε εκ του μηδενός την ανοικοδόμηση κάθε φορά. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Ίσως κάποια ασφαλιστικά προγράμματα. Ο ρόλος επίσης ε, του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντικός για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη. αλλά η Ένωση που είναι ένα σημαντικός χωρικός έχει επίσης το ρόλο της. Θα μπορούσα να πω και σε πιο μεγάλε λεπτομέρειες για την κατανομή ακριβώς της ε, βοήθειας που θα δεσμευτούμε να παράσχουμε σε περιφερειακό επίπεδο αν θέλετε. Αλλά θα σταματήσω εδώ κάνοντας απλά μια γενική επισκόπηση προ το παρόν τη υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μέσο μακροπρόθεσμη ανάκαμψη Τη περιοχή και την μεγαλύτερη τη ανθεκτικότητα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Αντέλβη, γιατί δεν ξέρω, φαντάζομαι ο κύριο Πόγκα θέλει το λόγο. Α, όχι, πρώτα ο Ενρικέ Γκερέρο. Συγγνώμη, εγώ τα μπέρδεψα. Ενρικέ Γκερέρο. Ήταν εκπρόσωπο ε, ο κύριο Ενρίκη και μόνιμο ηγητή για τα θέματα τη τροπιστική βοήθεια και αυτό έχει πρώτα τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ και του τρει σα για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για το πάθος με τον οποίο προσεγγίσατε το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ, χρησιμοποιώντας τα ισπανικά, υπάρχει ένα σύνολο καταστάσεων που ξεκινούν από «η». Ε, δεν μεταφράζεται φυσικά στα ελληνικά αυτά. Το γεγονός ότι συνέβησαν όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα, τα καταστροφικά, όπως είπε και η κυρία Κίμολ σε 15 μέρες είχατε δύο τυφώνες οι οποία ήταν η πιο καταστροφική σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο που αυτά το φετινό καλοκαίρι αποκλειστικά και μόνον. Διαπιστώνεται ότι ε, τα φυσικά φαινόμενα αυτά τα οποία ε, σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ε, τείνουν να επαναλαμβάνονται και επομένως ε, το αναμενόμενο θα είναι στο μέλλον να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ε, τέτοιων καταστροφών. Το δεύτερο είναι ότι είναι ε, αναπανόρθωτη ζημιά. Υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, πεθαίνουν, άνθρωποι θύματα αυτών των φυσικών καταστροφών και σε αυτή την περίπτωση επιπλέον και αναπανόρθωτη ε, η φυσική καταστροφή σε κάποιες κοινότητες τις οποίες η φύση είναι βασικός τρόπος επιβίωσης. Είναι αυτό το οποίο προσελκύει την οικονομική δραστηριότητα που επιτρέπει να επιβιώσετε. Και επομένω, ένα φαινόμενο αυτής της μορφής ε, δεν αφαιρεί μόνο ανθρώπινες ζωές, που σίγουρα είναι το χειρότερο απ' όλα, αλλά αφαιρεί και τον τρόπο ζωής αυτών των κοινοτήτων. Το τρίτο είναι η αδικία αδικία υπό την έννοια ότι όπως ε, αναφέρθηκε είστε θύματα ε, από φαινόμενα τα οποία προέκυψαν από τη συμπεριφορά άλλων χωρών, άλλων υπήρων που είναι πιο ανεπτυγμένε ή που είναι σε διαδικασία ανάπτυξης που εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερο ε, αριθμό αερίων που ε, λύνουν, ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα, που είναι υπεύθυνε για την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο και καταστρέφονται περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν λιγότερο σε αυτή την επιζήμια συμπεριφορά. Κατόπιν έχουμε και την αδυναμία να ανταποκριθούν αυτές οι κοινότητες μόνες τους ε, στα όσα προκύπτουν και ε, το θέμα της αλληλεγγύης ε, φυσικά. Το Κοινοβούλιο έστειλε αντιπροσωπεία στην συνεδρίαση στο Κανκούν της παγκόσμιας πλατφόρμας της ε, παρακολούθησης ε, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές ή καταστροφές άλλου τύπου και λίγους μήνες μετά πρώτα είχαμε το σεισμό στο Μεξικό και μετά του ε, τους τυφώνες στην περιοχή της Καραϊβικής και ε, Όλα αυτά κατέδειξαν και το πόσο απαραίτητα ήταν όλα όσα συζητήθηκαν στο Κανκούν. Στο Κανκούν, επειδή ε, προέκυψε και από τη ε, συμφωνία του Σεντάι, δύο διαφορετικές πτυχές. Η μία είναι σίγουρα η αλληλεγγύη ε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα φαινόμενα και μας είπαν ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει σήμερα δέσμευση για πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σίγουρα σημαντικό το ποσό, δεν επαρκεί για τις ζημίες που προκλήθηκαν, αλλά είναι σημαντικό ποσό και επομένω πρέπει να νιώσουμε και ικανοποιημένοι και περήφανοι για αυτή τη βοήθεια και την ένδειξη αλληλεγγύης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο οι στρατηγικές ε, προετοιμασίας ε, για τις φυσικές καταστροφές, ε, για να μπορούμε να απαντάμε σε αυτές τις φυσικές καταστροφές που ανέφερε και ακροθυγό στο τέλος της παρέμβασής της η κυρία Άντερσεν. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα τώρα, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι φαινόμενα ρουτίνας υπό την έννοια ότι επανεμφανίζονται κάθε χρόνο και επομένως ε, θα μπορούσαμε ίσως να είναι προβλέψιμα και να ε, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη τον ε, ε Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη των καταστραφών, τον κύριο Γκλέισερ, ε, μπορούν να ε, αναπτύξουν και να βοηθήσουν για την ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών για την προετοιμασία των χωρών της περιοχής. Βεβαίως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν θα επιληθούν ούτε με χρήματα ούτε με κατάλληλη προετοιμασία, αλλά ε, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας να επιδείξουμε αλληλεγγύη για την περιοχή, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πάντα θα είναι υπέρ της αύξησης της δυνατοτήτων αλληλεγγύης. Και ένα τελευταίο και νομίζω ότι αυτό ε, περιλαμβάνεται και ε, στο ζουμί ουσιαστικά της πρώτης παρέμβασης που ακούσαμε. Πρέπει να διευκολύνουμε την οικονομική δραστηριότητα, το εμπόριο με την περιοχή, με συμφωνίες ε, οικονομικής φύσεως, αλλά και με εμπορική συμπεριφορά, αν θέλετε, η οποία δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη της περιοχής. Ε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η φυσική καταστροφή είναι τόσο μεγάλη που η δυνατότητα ανάκαμψη είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά σύν το χρόνο θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ανάκαμψη και αυτή τη στιγμή ε, δεν αρκεί μόνο να σας υποστηρίξουμε με πόρους, αλλά και με ένδειξη αλληλεγγύης και μια ε, κατάλληλη εμπορική πολιτική και πολιτική ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο. Θα σας ζητήσω να είστε σύντομοι, 1,5 λεπτό ο καθένας, γιατί μετά θα πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα της ώρας των ερωτήσεων και έχουμε και τη συνάντηση των συντονιστών. Επομένως δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Κύριος Νόιζερ ξεκινάμε, ε, όχι, συγγνώμη, κύριος Πόγκα, Νόιζερ και τέλος τον Άνω. Συγγνώμη κυρία Ντονάνο, στον κύριο Πόγκα έδωσα το λόγο πρώτα. Ζητά συγγνώμη κυρία Ντονάνο. Κύριο Πόγκα. Σα ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο. Έχω δύο ερωτήσει. Αφού πρώτα βεβαίω ευχαριστήσω του τρει ομιλητέ που μας εξήγησαν την κατάσταση σε αυτά τα τρία μικρά νησιά μετά το χτύπημα των τυφώνων. Το πρώτο ερώτημα. Μιλήσατε για 300 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, συμπεριλαμβάνονται ε, στους ε, δωρητές, ε, μάλλον δεν συμπεριλάβατε στους δωρητές που αναφέρατε, τις χώρες της περιοχής της υπερπόντης κτήσης Σαμαχτά και η Ανγουίλα. Θα μπορούσαν και αυτές να επωφεληθούν από τη βοήθεια αυτή. Και το δεύτερο ερώτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής συγγνώμη, ε, ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Τι κάνετε για το, την σχέση μεταξύ Σαν Μαχτάν και Σαν Μαρτίν. Ε, τι, υπάρχει μια ξεχωριστή χρηματοδότηση για το Σαν Μαρτίν, προπόντια εκτίση της Ολλανδίας, ή για το Σαν Μαρτάν, προπόντια της Γαλλίας ή από κοινού, γιατί πλήγησαν και, και οι δύο αυτές περιοχές από τους ίδιους τυφώνες. Αυτές οι δύο ερωτήσεις από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Νόρμπερτ. Και από τη δική, τη δική μου πλευρά ευχαριστώ. Είμαι αριστερά μπροστά μπροστά. Ο Ενρίκε ουσιαστικά είπε τα πιο ουσιώδη, τα πιο βασικά. Πράγματι διατρέχουμε τον κίνδυνο να δούμε νησιά που στο μέλλον θα είναι σχεδόν ακατοίκητα. Γιατί έχουμε δραματικές κλιματικές αλλαγές. Εφόσον αυτό συνεχιστεί, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Πώς μπορούμε την ανθεκτικότητα των νησιών να την ε, βελτιώσουμε. Είπατε ότι υπάρχουν μέσα και υπάρχει και διμερός ε, και πολυμερός η δυνατότητα παροχής βοήθειας και ενίσχυσης. Εδώ, στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, έχουμε πάρει κονδύλια τούτο. Είναι διαθέσιμα κονδύλια και είναι και βιώσιμος ο σχετικός σχεδιασμός. Και μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το κατά πόσο υπάρχουν διαφορές ε, στη βοήθεια που έχει να κάνει με τα, την Ανατολική, Καραϊβική, την Κούβα και άλλες περιοχές, γιατί με την Κούβα νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Και το άλλο θέμα που το ανέφερε και ο Ενρίκε, αλληλεγγύη δείχνουμε ένα μικρό παράδειγμα αλληλεγγύης. Η επόμενη ισομερής ε, ε, συνέλευση θα γίνει στην ΑΕΤ. Ε, μιλάω για την ισομερή συνέλευση και εκπροσώπησης χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέλλον νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εντατικοποιήσουμε τη βοήθεια να αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία. Τώρα. Ρε κυρία Τορνάνο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα επανέλθω στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Πόγκα. Πράγματι, έχουμε δύο περιοχές που, κατε, που Σαν Μαχτάν και Σαν Ματίν, 80% του εδάφους έχει καταστραφεί. Ε, πρόκειται για εξαιρετικά απόμακρες περιοχές και είχαμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα σε ε, χιλιάδες ε, κατοικίες. Στη Μαρτινίκ χάσανε όλη την σοδιά μπανάνας που είναι η πιο σημαντική πηγή ε, της αγροτικής οικονομίας. Η Γαλλία έχει αναλάβει πρωτοβουλία βεβαίως για να βοηθήσει τις ε, περιοχές αυτές αλλά ε, δεν επαρκεί. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει κρατήσει 95 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά χρειάζεται και η διεθνής βοήθεια, η διεθνής αλληλεγγύη και όχι μόνο για την άμεση ανταπόκριση, αλλά και για το μετέπειτα, για την, την πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Τι λοιπόν προβλέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσει τις περιοχές αυτές τις γαλλικές, την αλληλεία, τον τουρισμό, την γεωργία, τομείς δηλαδή της οικονομίας οι οποίοι επλήγησαν και, θα πρέ... και για τις οποίες, και για να βοηθήσουμε τους... αυτούς τους τομείς, ε, θα πρέπει να κατατήσουμε ένα γενικότερο και πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο απαντήσεις, αλλά με την αντίθετη σειρά. Πρώτα ντεύκο, γιατί νομίζω ότι είναι ορισμένα ερωτήματα για εσάς, μετά έκο και στο τέλος η κυρία Μακλίνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας, κυρία Αντρίανσεν. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα κατά πόσον ε, καλύπτονται άκρως από κέντρες περιφέρειες και τα ντομ-τομ, ε, ε, περιοχές εδάφη. Ξέρετε ότι έχουν διαφορετικό καθεστώς. Σε ό,τι αφορά τις άκρως από κέντρες ε, περιοχές υπάρχουν διαφορετικά πλαίσια υποστήριξης ανάλογα με την περιφερειακή πολιτική. δεν μπορώ εγώ να σα επιβεβαιώσω για την άλλη αρμόδια γενική διεύθυνση σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει αυτέ τι εξόχως περιοχέ. Ε, περιοχές. Για τα περπόντα εδάφη που εντάσσονται ή καλύπτονται τέλο πάντων από το ΕΤΑ, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι θα τα στηρίξουμε απάντα και του κ. Πόγκα εφόσον έχουν πληγεί από τους άσφατους αυτούς τυφώνες. Προς το παρόν περιμένουμε ακόμη να ολοκληρωθούν αξιολογήσεις μετά τις καταστροφές αυτές για να επιβεβαιωθεί το εύρος η έκταξη των ζημιών και να προσδιορίσουμε τα ποσά τα οποία θα χρειαστεί να δοθούν. Έχουμε όμω ήδη βάλει στην άκρη ένα αποθεματικό για να καλύψουμε τι ανάγκε αυτών των περιοχών. Υπάρχουν συνάδελφοι στην αίθουσα που εργάζονται στο θέμα αυτό πιο συγκεκριμένα. Αν έχουν να προσθέσουν κάτι καινούργιο, λέει πρόεδρο, ναι, να του δώσουμε το λόγο. Έχετε κάποια πληροφορία συγκεκριμένη. Αν όχι, δεν πειράζει. Μπορείτε να απαντήσετε γραπτό αργότερα. Μόνο αν έχετε νέε πληροφορίε. Ναι, ευχαριστώ κύριε. Πυρκίν. Πράγματι, για να απαντήσω συμπληρωματικά στα όσα ήδη δόθηκαν ως απάντηση στον κύριο Πόγκα για τα κοντήλια, 300 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια λίγο πολύ θα πάνε ειδικά στα βέρποντε εδάφη εφόσον έχουμε πάρει από τα κράτη αυτά συγκεκριμένα αιτήματα χρηματοδότησης για την κατηγορία Β. Πολλά εδάφη τέτοια έχουν πληγεί. Πήραμε ήδη έτοιμα από την Άγγελα για το εκπαιδευτικό σύστημα και περιμένουμε από το Σε και από τα Κάικος που θα υποβάλουν προτάσεις για τη διαφορά στο στάτους που είναι και το ένα ερώτημα για την έννοια για το Σερ Μαρτέν και το Σερ Μαρτίν. Το ένα είναι άκρος από κεντρική περιοχή, το άλλο είναι υπερπόντιο διαμέρισμα. Δεν είναι η ίδια μεταχείριση. Βέβαια, Ήδη υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν την ε, κινητοποίηση πόρων ε, για το Σεν Μαρτίν, το υπερπόντεο διαμέρισμα που κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσουμε από κοινού το Ταμείο Ίντερεκ ε, και το ΕΤΑ. Με το Ίντερεκ μπορούμε να έχουμε γέφυρες μεταξύ των δύο χρηματοδοτήσεων. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και θέλουμε να ενθαρρύνουμε αυτού του είδους τη συνεργασία. Το έχει επιβεβαιώσει και σε απάντηση του στον κύριο Ταγιάννη ο πρόεδρος της Κομισιόν, κύριος Γιούγκερ. Ο κύριος Λάνσκραφ έχει να προσθέσει κάτι μήπως. Ευχαριστώ πολύ σύντομα για να απαντήσω στον κύριο Γκερέρο και στον κύριο Νόιζερ. Ναι, νομίζω ότι από όλες τις ενδείξεις που έχουμε, η κλιματική αλλαγή είναι ένας ακόμα παρόγων που ε, αυξάνει την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια παγκοσμίω και πράγματι συμφωνούμε και εμείς ότι πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε ε, ε, ποσά και να προσέχουμε ιδιαίτερα την προετοιμασία για τις καταστροφές. Έχουμε μια ιστορία άνω των 20 χρόνων σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο συνέβαλε και στην Καραϊβική όπου πραγματικά χρειαζόμαστε να δούμε ε, συγκεκριμένες δυνατότητες ε, για τη μείωση ε, των καταστροφών και την προετοιμασία των καταστροφών. Και αυτό έχει αποδειχθεί όχι μόνο από τις παρεμβάσεις του συντήμα και το, η στήριξη και των παρεμβάσεων σε κάθε χρόνο ε, κάθε χώρα συγγνώμη, υπάρχει ε, συγκεκριμένος βαθμός προετοιμασίας για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί. Επίσης, πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε και καινοτόμα προγράμματα, όπως για παράδειγμα ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία θα μπορούσαμε να χρηματοδοτούσαμε με συμπράξη δημοσίου ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και μια σύντομη απάντηση και στον κύριο Πονγκά. Ε, ίσως ε, παρανόησα, δεν ήταν 300 εκατομμύρια, μακάρι να είχαμε τόσο λεφτά για αυτή την απάντηση. Ε, κάτι σε 3 εκατομμύρια ευρώ έχουμε για ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό έχει παρασχεθεί. Και όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια ε, για τις υπερπόντιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερθήκατε στη Μαρτινίκα, στη Γουαδελούπη και στο Σαμαρτά ε, και εσείς κυρία Τορνανό, ε, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη νομική βάση δεν μας επιτρέπει να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ε, μπορούμε να παρέμβουμε στο Σαν Μάρτιν, όπου δώσαμε βοήθεια για στέγαση, αλλά όχι για το Σαν Μαρτάν, γιατί είναι υπερπόντια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα ανθρωπιστικά ε, θέματα λοιπόν είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Τα ανέφερα λοιπόν και ε, συγγνώμη αν δεν ανέφερα τα πάντα, Αντίγουα, Μπαρμπούντα, Κούβα και Δομίνικα ανέφερα. Αλλά επίσης και στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην Αϊτή, στο Σαν Νέβης και στο Σαν Μάρτιν που μόλις ανέφερα ε, και στα Κάικος ε, Έλα δόθηκε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τέλος η κυρία ε, Σίλιφεν δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, πολύ σύντομα. Ε, καταλαβαίνω ότι σας πιέζει και ο χρόνο. Να πω απλώς ότι στην περίπτωση της ε, Δομίνικα και της Αντίγουα οι αξιολογήσεις ε, των αναγκών μετά την καταστροφή κατέδειξαν ότι ε, βάσει της έκθεσης της Παγκόσμιας Παρ, ε, Τράπεζας των Ηνωμένων ε, Εθνών κλπ. έχει πάνω από 3 δις ε, δολάρια ζημιά που είναι περίπου το 30% του ΑΕΠ. Μέσα σε 46 ώρες η Αντίγκουα και η Μπαρμπούντα καταστράφηκε ολοσχερός και έχουμε 400 εκατομμύρια ζημιά. Αυτό λοιπόν βιώνουμε αυτή τη στιγμή και σίγουρα η βοήθεια και η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ανθρωπιστικό επίπεδο αλλά και μακροπρόθεσμα μέσω της διάσκεψης των δωρητών ε, ε, την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Όπως διαπιστώνετε θα είναι απλώς τμήμα των όσων χρειαζόμαστε αλλά είναι τόσα πολλά πράγματα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Και να περάσω πολύ γρήγορα στα πρώτα σχόλια που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον και να σας πω ότι ε, Γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιος βαθμός προετοιμασίας, έχουμε εμπειρία με τυφώνες, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να μας είχε προετοιμάσει για δύο τυφώνες κατηγορίας 5. Και η καταστροφή και των υποδομών είναι ε, πολύ σημαντικό ζήτημα. Και θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα και στο δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι ε, ως Καραϊβική αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα την όλη συζήτηση για τη νομική βάση που έκαναν οι συνάδελφοι σας και αυτό είναι περίεργο, διότι ο άνεμος δεν ξέρει τίποτα για αυτά τα όρια και ο άνεμος δεν γνωρίζει τίποτα για τις νομικές συμφωνίες ε, ε, που θεωρούν το Σαν Μαρτάν διαφορετικό από το Σαν Μάρτιν. Ε, και πρέπει να σας πω ότι η οικογένειά μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη Μαρτινίκα και ε, πήγανε στη Μαρτινίκα, από τη Μαρτινίκα στη Δομίνικα ε, το 1979 έγινε ένας τυφώνας που κατέστρεψε τη Δομήνικα και η μισή μου οικογένεια γιατί ήταν Γάλλοι, είχαν δικαίωμα και έφυγαν. Όποιο δεν είχε τέτοιο δικαίωμα έμεινε. Ο άνεμος λοιπόν δεν τα γνωρίζει όλα αυτά τα νομικήστικα και τα σύνορα και τα τερτύπια του νόμου. Και για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μακροπρόθεσμα να δούμε τι συμβαίνει στο Βόρειο Ατλαντικό με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Πραγματικά πρέπει να εξετάσουμε τις χώρες και τις νήσους ε, του Βορείου Ατλαντικού ως ε, ανθρώπους που βρίσκονται στις παρυφές. Ε, ε, είμαστε στις παρυφές λόγω των, της εθνικότητάς μας, της ηθαγένειάς μας, της τοποθεσίας μας. Είμαστε μικροί και βάλωτε. Και είναι πολύ δύσκολο να αιτιολογήσουμε τη βοήθεια και την ανάγκη για βοήθεια. Όσο και αυστηρή να είναι νομική βάση, είναι δύσκολο να αιτιολογήσει κάποιο γιατί θα βοηθήσει μισό νησί και όχι το άλλο μισό. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνουν όλοι αυτοί που έχουν την εξουσία και φυσικά αυτό δεν είναι στα χέρια των χωρών αυτών της καρεβική. Πρέπει να δείτε αυτό που ζητάμε. Ζητάμε να υπάρχουν κάποια μέσα, κάποια κατηγορία ταμείου που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσω και θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε χώρε οι οποίε πλήττονται από τέτοιε καταστροφέ. Και αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ε, ευρωπαϊκή επικράτεια, υπερπόντια εδάφη, ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε, γιατί είμαστε όλοι μια οικογένεια. Παντού χάνονται ζωέ όσε χάθηκαν στη Μαρτινίκα, χάθηκαν και στη Δομήνικα και στο Σαμαρτάν και στι βρετανικέ Παρθένε νήσου έχουμε στενές σχέσεις, είναι τμήμα της κληρονομιάς μας και υποφέρουμε και από κοινού. Αυτή λοιπόν είναι μια τελευταία σκέψη. Πρέπει να γίνει αυτό μακροπρόθεσμα και πρέπει να επιδείξουμε καινοτιμία. Πρέπει να σκεφτούμε νέα μέσα, να κάνουμε κάτι γιατί δεν αρκεί τα, ο, ο status quo. Δεν αρκεί. Ε, και στα ισπανικά το είπε ο Μιλήτρη. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνετε, ότι προφανώ δεν γνωρίζουν οι φυσικέ καταστροφέ ούτε τα σύνορά μα ούτε τα Brexit μα ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο ήρθε και επανήλθε στη σημερινή συζήτηση ε, όταν έχουμε τέτοιου είδου φυσικέ καταστροφέ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα, για την παρουσία ε, εδώ και τι παρουσιάσει σα ελπίζουμε και θα σας προσκαλέσουμε να επανέλθετε στην Επιτροπή μας για να μας ενημερώσετε για την πορεία ε, της αντιμετώπισης αυτής της καταστροφής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε γρήγορα στην ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή μας. Είναι το τελευταίο, πρώτο τελευταίο μάλλον σημείο της ημερησίας μας διάταξης με δύο ερωτήσεις από την κυρία Σαρτζεντίνη Πρώτα είναι η διαδικασία του Κίμπερλι για την πιστοποίηση των διαματιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει, αν δεν απατώμε την επόμενη χρονιά, την ηγεσία αυτής της, ε, αυτού του οργανισμού, της διαδικασίας του Κίμπερλι και ε, το ερώτημα απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα, τα βασικά, σας παρακαλώ μόνο να μας ενημερώσετε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε διευθύντρια της υπηρεσίας που ασχολείται με ε, εργαλεία εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα επαναλάβω αυτό που είπατε. η διαδικασία του Κίμπερλι είναι μια πρωτοβουλία διεθνής για, την προστα... για ε, να σταματήσει το εμπόριο των λεγόμενων ματωμένων διαμαντιών, ε, διαμαντιών που έχουν προέλθει από περιοχές συγκρούσεων. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2003, ε, στην οποία συμμετείχαν πολλές χώρες από τι οποίε εξάγονται διαμάντια, συμπεριλαμβανομένες και τη νότια Αφρική. Ε, αυτή τη στιγμή την Προεδρία έχει η Αυστραλία, από την επόμενη χρονιά θα την αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε τρία χρόνια γίνεται μια αξιολόγηση για να δούμε πώς λειτουργεί η διαδικασία. Ο τρέχον προγραμματικό κύκλο έχει ξεκινήσει φέτο και θα συνεχίσει του χρόνου. Ε, εξετάζουμε ζητήματα όπω η διαδικασία λήψη αποφάσεων και πώ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική. Η διαδικασία τη αξιολόγηση από ομότιμα μέρη. Ε, ο ορισμό του τι συνιστά εμπολεμιζών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιοποιήσει την Προεδρία της για να προωθήσει τη χρήση αυτής της διαδικασίας και να δει πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερο συντονισμός με άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας των φυσικών πόρων και της δίωσης επιμέλειας όταν χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι από οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου. Οι αποφάσεις στη διαδικασία του Κίμπελ λαμβάνονται με ομοφωνία. Επομένω πρέπει να υπάρχει συμφωνία όλων πριν οποιοδήποτε αλλαγή γίνει στην πράξη. Από την πλευρά τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τέσσερι προτεραιότητε κατά τη διάρκεια τη προεδρία τη. Πρώτον, να ενισχυθούν οι τρεις, η σχέση μεταξύ των τριών ε, πυλώνων, των τριών συμμετέχοντων, συμμετεχόντων μερών στην διαδικασία του Κίμπελη, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις. Μετά να βελτιωθεί το σύστημα της πιστοποίησης με ανταλλαγή των βελτιστών πρακτικών, με την συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην εφαρμογή των πιστοποιητικών, τη δίωξη δηλαδή αυτών που τον παραβιάζουν. Αυτό θα γίνει με καλύτερη ανταλλαγή των πληροφοριών και ενθαρρύνοντας την συνεργασία ε, μεταξύ της συμμετοχόντων για να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο των πολύτιμων λίθων και να υπάρχει καλύτερη αστυνομική συνεργασία. Αυτή ήταν η δεύτερη προτεραιότητα. Η τρίτη προτεραιότητα είναι ε, η βελτίωση των δυνατοτήτων ε, των κρατικών αρχών και να δούμε πώς η διαδικασία του Κιμπερλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να, πάμε προς, ε, να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης <clears throat> και των σχετικών συμβάσεων του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου φυσικών πόρων. Θα δούμε ποιες χώρες χρειάζονται τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα, τέτοια προγράμματα κατάρτισης και τι μπορούμε να κάνουμε. Η τέταρτη προτεραιότητα είναι μια προτεραιότητα συνολικής ε, γενική και είναι η εξή, ότι, ότι σε οποιαδήποτε τη δραστηριότητα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια τη Πρωτοεδρία, θα αναδείξει το ζήτημα τη ισότητα των δύο φύλων και τη προστασία των παιδιών. Αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία ε, με τα οποία θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα τη Επιτροπή σα και ευχαρίστω να απαντήσω, να σα δώσω περισσότερε πληροφορίε αν το επιθυμείτε. Κυρία Σαρτζεντίνη, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, τη γνωρίζω πολύ καλά τη διαδικασία Κίμπερλι, λοιπόν, ξεκίνησε και μάλιστα ήμουν και στις τριμερείς διαπραγματεύσεις ε, ως εκπρόσωπος της κοινωνία των πολιτών μεταξύ του 2000 και 2003, οπότε και διαπραγματευθήκαμε την εν λόγω νομοθεσία. Και εξακολουθώ να νιώθω ευγνωμοσύνη προς την Κομισιόν που ήταν κινητήρος μοχλός τότε από τη στιγμή που θα έχετε προεδρία του χρόνου, του παραχρόνου, σημαίνει τώρα έχετε την αντιπροεδρία. Έτσι τουλάχιστον λειτουργούσε το σύστημα. Άκουσα τις τέσσερι προτεραιότητές σα. Γνωρίζουμε όμως και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα με την νομιμοποίηση της διαδικασίας Κίμπερλι και το πρόγραμμα πιστοποίηση. Γίνονται καταχρήσεις ό,τι αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το πρόγραμμα όμως επισήμως ε, το ορίζουν οι χώρες που δεν βλέπουν τις καταχρήσεις που γίνονται από τις χώρες, αλλά καταχρήσεις που γίνονται από ομάδες επαναστατών. Είδαμε κάποια σκάνδαλα όμως, ε, ένα στην Νότια στη Ζιμπάμπου η κατάσταση, οι κυβερνήσεις εποφελούνταν και παρατηρείται καταχρήσεις και καταπατήσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαδικασία Κίμπερλι πολύ αγρά, αργά αντιδρούσε στις προκειμένες αυτές περιπτώσεις. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται με τα ορυχεία και ιδίω με τις γυναίκες και τα παιδιά. Για να είναι μια σεβαστή διαδικασία αυτή, η διαδικασία Κίμπερλι, Ίσως του χρόνου ως πρόεδρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναζητήσει όχι μόνο τη συνένεση, γιατί με χώρες όπως τη Ζιμπάμπου δεν είναι και τόσο εύκολο να αναζητεί κανεί συνένεση. Θα πρέπει όμως να δραστηριοποιηθεί εκ των προτέρων για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παραβίασης των δικαιωμάτων και από μέλη της διαδικασίας Κίμπερντ, η Κομισιόν. Καλή είναι η απάντησή σας, είναι όμως κάπως γραφειοκρατική. Ευχαριστώ. Hey. Thank anything η Κομισιόν πως θέλει κάτι να προσθέσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Σαρτζεντίνη. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαστε κάθε άλλο παρά κρατική όσο θα έχουμε την Προεδρία. Τώρα, ότι... δηλαδή θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που θα μας δοθεί για να θέτουμε αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε. Βέβαια ταυτόχρονα θα πρέπει να εργαστούμε και στο πλαίσιο που ορίζεται από τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα ματωμένα διαμάντια και τον ορισμό αυτών των πολύτιμων λίθων από περιοχέ τη σύγκρουση. Νομίζω ότι είναι προ όφελο όλων των συμμετεχόντων, όπω είπατε, η διαδικασία να παραμείνει προσαρμοσμένη στο σκοπό που θέλει να υπηρετήσει και πρέπει να είναι πιο ευρύ ορισμό ε, ε, αυτών των conflict diamonds για να ανταποκρίνεται στο τι γίνεται επί τόπου. Το 2012 η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε τη διεύρυνση του, της εντολής, ώστε η διαδικασία να μπορεί να αντιμετωπίζει ευρύτερες ε, περιπτώσεις ε, συγκρούσεων, παραβιάσεων και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2018 ως Προεδρία θα διευκολύνουμε τη διαδικασία και τη συζήτηση για ενδεχόμενη διεύρυνση της εντολής. Όπως είπα, χρειάζεται συνένεση όμως για την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Προεδρία. Επειδή έχουμε πρόσβαση στις συμμετέχουσες χώρους και έχουμε επαφές για να επηρεάσουμε για την ε, παροχή βοήθειας. Να θέσουμε τον δάκτυο από τον τύπο των ήλων, όπως είπατε, να ζητήσουμε την προσοχή τους και να έχουμε θεταμένες συζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερο με τις συμμετέχουσες χώρες. Η διαδικασία Κίμπερλι θα πρέπει να δοθεί συμπληρωματικά και προ τη διαδικασία τη δέωση επιμέλεια ή των προσπαθειών που γίνονται είτε στον ΩΣΑ είτε σε διεθνή φόρα όπω η Διεθνή Οργάνωση Εργασία των ΗΠΑ. Εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε συνέργειες με άλλου διεθνεί οργανισμούς και πρωτοβουλίε όπου αυτό είναι δυνατόν και έχει σημασία. Στο πλαίσιο τη επερχόμενη Προεδρία μα. Δεν μπορώ βέβαια να σας υποσχεθώ ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τον ορισμό. Μπορώ να σας υποσχεθώ όμω ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσελκύσουμε την προσοχή στο θέμα και θα αξιοποιήσουμε τις επαφές μας για να θέσουμε αυτό το ζήτημα και για να μετακινηθούν οι κυβερνήσει και οι άλλοι φορείς. σε ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Και εγώ ήμουν εδώ όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία και θέλουμε να πετύχει γιατί θέλουμε να αυστηροποιήσουμε και κάποιες άλλες κατευθύνσεις γραμμέ του ΟΣΑ. Και αν δεν το καταφέρουμε εδώ, δεν θα το καταφέρουμε και με άλλε. Ένα άλλο ερώτημα της κυρίας Αργεντίνη αφορά την Επιτροπή ΝΤΑΚ του ΩΣΑ και τη συμμετοχή της Κομισιόν. Θέλουμε να ενημερώνεται η Επιτροπή μας περισσότερο για το τι συμβαίνει, για το τι λέγεται στις συναντήσεις ψηλού επίπεδου ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκπρόσωπο της Ένωσης. Δεν ξέρω ποιον έχουμε εδώ από την Κομισιόν θα απαντήσει το ερώτημα αυτό. Εσείς παρακαλώ. Δεν έχω το όνομά σας, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νικολέτα Μέρλα, αναπληρώτρια τμήματάρχης ε, στο τμήμα χρηματοδότησης και αποτελεσματικότητας της ΔΕΒΚΟ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση μετά από την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου. Αυτή η 51η συνεδρία σε υψηλό επίπεδο έγινε στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο Παρίσι και ο στόχος ήταν να εγκριθεί η νέα εντολή και η νέα στρατηγική για την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τη νέα αναπτυξιακή αρχιτεκτονική, το θεματολόγιο του 2030 και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης στόχο είχε να ολοκληρώσει τη διαδικασία του εξυγχρονισμού που ξεκίνησε το 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Στέφανο Μανσερβίζη, το Γενικό Διευθυντή της της ΔΕΒΚΟ. Η συνεδρίαση υψηλού επίπεδου ενέκρινε τις διευκρινήσεις ε, στην στατιστική ε, ε, στις εκθέσεις μάλλον των στατιστικών των χωρών δωρητών και αυτό είναι αποτέλεσμα εργασιών που έγιναν ε, σε μια προσωρινή ομάδα εργασίας η οποία συστήθηκε το Φεβρουάριο και ο στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να υπάρξουν διευκρινήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των εκθέσεων που υποβάλλονται από τα μέλη της ΔΑΚ. Βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποβάλλει εκθέσεις ε, στο ε, στα θέματα αυτά, αλλά ε, θεωρεί την πρόταση ευπρόσδεκτη γιατί αυξάνει την ε, συνέπεια και την ευθυγράμμιση με την οποία υπολογίζεται το κόστος για τους πρόσφυγες μεταξύ των χωρών. Δεν υπάρχει επέκταση του πεδίου εφαρμογή των ε, υποχρεώσεων υποβολή έκθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θετική στάση για αυτή την πρόταση, την οποία βρήκε ιδιαίτερα ισορροπημένη. Όπω γνωρίζετε, βεβαίω από εκεί και πέρα έχουμε ένα ρόλο γιατί μπορούμε να ε, ε, εδραιώσουμε τη θέση των κρατών μελών και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέπεια των εκθέσεων συνολικά. Όσον αφορά το θεματολόγιο της ε, συνεδρίασης υψηλού επίπεδου υπήρχε και το θέμα των ε, λεπτομεριών για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων. Είναι μια πρόταση η οποία ήρθε μετά από μια αρκετά μακρά διαδικασία, μια πρόταση να μεταφραστούν οι αρχές για τον εξυγχρονισμό για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα που εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση υψηλού επίπεδου το 2016 και πρότειναν αλλαγή από εκθέσεις ε, για τη ροή μετρητών, ε, για να αναφέρονται από τη μια η οριμότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται, αλλά και το επίπεδο κινδύνων και το ε, επίπεδο των άλλων χωρών. Η πρόταση αυτή ε, κατά την Επιτροπή ήταν ισορροπημένη και συνάδει και με τις απαιτήσεις ε, της ατζέντα δράση τη Αντισεβέμπα που ε, περιλαμβάνει και τη δέσμευση να υπάρχει και μόχλευση των πόρων του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των υποδομών και ε, περιλαμβάνει και την αναγνώριση κάποιες από τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων και το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που εγκρίθηκε. Ε, Δυστυχώ ε, δεν εγκρίθηκε από όλα τα μέλη της ΔΑΚ, επομένως δεν εγκρίθηκε η πρόταση αυτή. Επομένως, ε, προς το παρόν θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε στην υποβολή των εκθέσεων για αυτές τις δραστηριότητες τις οδηγίες του 2012 που ακόμα διατηρούν μια προσέγγιση όσον αφορά τη ροή μετρητών και δεν περιλαμβάνουν και τις εγγυήσει εκτός και αν ενεργοποιηθούν. αυτά λοιπόν εν είδη ενημέρωσης σε απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Αρζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Τζούντιφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συνάδελφος η Μαρία Χόιμπουχ έθεσε ερωτήσεις στις 10 Οκτωβρίου για την προετοιμασία αυτής της συνεδρίας υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι είχαμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΔΑΚ που ήρθε εδώ νωρίτερα όταν συζητήσαμε τις αλλαγές ε, στα κριτήρια του ΝΤΑΚ και πιο συγκεκριμένα τη μετανάστευση και νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς προσπαθούμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει και λίγο καλύτερα και ποιος παρέχει την εντολή για να βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί και να λαμβάνει αποφάσεις. Ε, αν η εκπρόσωπο της Επιτροπής αναφέρει τις προτάσεις που ετέθησαν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εμείς ακόμα δεν τι έχουμε δει τις προτάσεις και νομίζω ότι καλό θα ήταν να δούμε προτάσεις ε, σαν αυτές, διότι όταν μου λέτε ότι είναι καλή ή δεν είναι καλή, αλλά εγώ δεν μπορώ να την αξιολογήσω γιατί δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται, δεν νομίζω ότι με βοηθά να προχωρήσω και να προσπαθήσω να καταλάβω την εντολή και τι πρέπει να γίνει από εκεί και πέρα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι κατά πόσον μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας αυτές τις προτάσεις ή τουλάχιστον τα αποτελέσματα των συζητήσεων μαζί μας και να μας πείτε περισσότερα και όχι απλώς ε, να μας τα λέτε προφορικά ε, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ε, διότι ε, υπάρχει και αξιολόγηση ισοτήμων από την Νορβηγία και την Ιαπωνία φέτο ε, για την βοήθεια που παρέχουμε. Και θα ήθελα να ξέρω αν έχει να διδραματίσει και κάποιο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την αξιολόγηση, διότι έχουμε και ελεγκτικό ρόλο για το αναπτυξιακή βοήθεια που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και θα ήθελα λοιπόν να θέσω την ερώτηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και σε εμά, κυρία Πρόεδρε. Τι ρόλο έχουμε όσον αφορά αυτή την αξιολόγηση ισοτήμων της Επιτροπής ΔΑΚ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το ελέγχω. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι μας είχαν αποστείλει τα έγγραφα για αυτή τη συνεδρίαση ε, πριν, ε, εγκαίρως, γιατί το είχαμε ζητήσει την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη μας συνεδρίαση. Τώρα βέβαια πρέπει να το ελέγξουμε, πρέπει να ελέγξουμε τα email, λαμβάνουμε εκατοντάδε την ημέρα. Ε, δεν θυμάμαι τώρα βέβαια αν τα λάβαμε τα έγγραφα πριν ή μετά τη συνάντηση. Πάντω σε κάθε περίπτωση μπορεί να βελτιωθεί. Ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία, μια γραπτή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του ζητήματο αυτού, αφού από την πλευρά τη λέει ότι δεν έχει καμιά αντίρρηση να ε, μοιράζεται αυτέ τι πληροφορίε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο συστηματικά, ε, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι για αυτέ τι συζητήσει που γίνονται σε αυτή την Επιτροπή ε, και να μπορούμε να τι παρακολουθούμε. Εντάξει, Judith. Ναι. Δεν έχουμε κανένα σημείο επί τα διάφορα. Η επόμενη μας τακτική συνεδρίαση θα γίνει στι 4 Δεκεμβρίου 2017, 3 η ώρα. Συνεχίζουμε με την συνάντηση των συντονιστών. Θα παρακαλέσω γενικά όλους όσους δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην αίθουσα να αποχωρήσουν. Καλό απόγευμα.